Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στην τρίτη ενότητα της συνεδρίασής μας. Και μεταδίδεται και στο διαδίκτυο όλη την ημέρα. Καλωσορίζουμε τους πρωινούς μας ακροατές um, και τηλεθεατές. Αρχίζουμε με μία ακόμα γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και μάλιστα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που κάνουν εκείνοι για το εμπόριο με την Κίνα. Είναι κάπως ε, επίμαχος και ο τίτλος. Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα, ε, έλλειψη ισορροπίας στο εμπόριο, ερωτηματικό. Να δούμε τι θα μας πει ο συντάκτης γνωμοδότησης, ο οποίος βιάζεται γιατί ξέρω ότι θέλει να φύγει να μην χάσει το τρένο του. Να του δώσω το λόγο. Δεν ξέρω πόσοι σκιώδεις είναι ε, παρόντες. Από τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι η κυρία Σαναλόβα. Αλλά η κυρία Σαλτεμόζε θα αναλάβει ε, την εκπροσωπήση. Η κυρία Ρούιλε νομίζω από τους Πρασίνου. Εγώ καλύπτω την κυρία <laughs> Μακλάρκιν που είναι στο Λονδίνο. Αλλά καλωσορίζω τον κύριο Τριανταφυλλίδη και χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να μας πει ε, για να μας εξηγήσει τη γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τους παρόντες που ήρθατε. Λέει ο κύριος Λόκεγκαρτ. Δεν μου αρέσει αυτό το ερωτηματικό κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνα μια εμπορική ανισορροπία λέει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που μας απασχολεί και δεν ξέρω αν θα πρέπει να το προεξοφλούμε. Είναι και νέα αρμοδιότητα για την Επιτροπή μας. Για το θέμα είμαι πολύ ενθουσιασμένος ε, γιατί είναι αρκετά ευρύ και έχουμε και μια ευκαιρία να ε, βρούμε κάποιες προτεραιότητες. Ήδη από χτε έχω πει ότι ισχύει για όλες τις εκθέσεις. Εγώ προσπαθώ να βρω μια ισορροπία με τη γνωμοδότηση. Τα τελευταία δέκα χρόνια ανοίγει η αγορά της Κίνας από την εισδοχή της στον ΠΟΕ και μετά. Αλλά πολλές φορές έχουμε ζητήματα κρατικών ενισχύσεων ε, ε, της κίνα, στις εταιρείε τους και άλλα κρυφά εμπόδια και φραγμούς ε, στο εμπόριο. Αυτή η ε, ανισορροπία υπάρχει, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κάνει η Κίνα, αλλά και τη δική μας στεναρή αντιμετώπιση των ε, φραγμών αυτών και της άρσης τους. Είναι ευαίσθητα θέματα αυτά, τα εμπορικά συνδέονται με νέες αρμοδιότητες για μας και πριν εμείς θα πρέπει να βρούμε ως Επιτροπή τη θέση μας εκεί. Είναι αρκετά άμεση η διατύπωση ε, στη γνωμοδότηση θα δείτε και εσκεμένα το έχω πράξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ε, με σαφήνεια. Ήδη από χτες και σημείωσα πρόεδρε ότι είναι κρίσιμο το θέμα και δεν θα πρέπει να το αφήνουμε μόνο στα χέρια των διπλωματών, αλλά να ασχολούνται και οι ειδικοί και πυρογνώμονες με φραγμούς εμπορικούς. Ε, είπατε ότι κάποιος ανέφερε ότι είμαστε ηγετική δύναμη στην τεχνολογία της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά θεωρώ φυσική τη δική μας συμμετοχή και τη σαφή μας θέση. Δύο λόγια για τη συνένεση και μάλλον για το ε, περιεχόμενο, την ουσία. Ε, το, η παράγραφος αναφερόνεται στο να εξηγεί τη, το τίτλο. Κάπου αναφέρεται τελικά η Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου με την Κίνα. Ε, γίνονται συζητήσεις με συμβούλους και εμπειρογνώμονες για αυτό το θέμα. Τελικά επέλεξα όμως να το αναφέρω παρόλα αυτά στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχουμε δύο φορές ετησίως ε, συνεδριάσεις με την Κίνα και όχι άπαξ. Και τα σημαντικότερα ζητήματα ε, είναι στο τέλος παραγράφου 2. Παράγραφος 3 έως 6. Περιγράφουμε περισσότερες λεπτομέρειες στα θέματα που μας απασχολούν. Η σειρά ε, με την οποία αναφέρονται δεν είναι τυχαία. Εγώ προτείνω να θέσουμε έτσι αυτές τις προτεραιότητες με αυτή τη σειρά. Είχα και επικοινωνία και επαφές με ε, διάφορους επιρρογνώμονες πριν γράψω τη γνωμοδότησή μου. Όπως είπα και στην αρχή, ένας συγγητής καλείται να κάνει δύσκολες επιλογές, γιατί έχουμε περιορισμένο χώρο. Καταλαβαίνω ότι θα γίνουν και πολλές τροπολογίες. Έχω και εγώ δικές μου, μεταξύ άλλων ε, μία για τις ε, πρώτες σύλλες ε, που δεν κατάφερα να τις χωρέσω στη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να σταματήσω εδώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εγώ προσωπικά δεν έχω χρόνο. Περιμένω τη δική σας συνεισφορά. Ο κύριος Κρόιτσμαν θα αναλάβει από εδώ και πέρα και είμαι βέβαιος ότι θα κάνει καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ευθεία η ε, γνωμοδότησή σας και πολύ καλά δομημένη. Μπορεί ορισμένοι να διαφωνήσουν, αλλά είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, ακόμα και αν χρειαστεί να φύγετε, θα σας ενημερώσουν. Ε, λοιπόν, ακούμε τους σκιώδεις ηγητές. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απουσιάζουν πάντα. Η κυρία Σάλντε Μόζε είναι έτοιμη να μιλήσει ε, από την ομάδα της. Ευχαριστώ. Ακόμα και αν έγινε πολύ ωραία συζήτηση Εχθές μιλούσα αγγλικά, σήμερα θα μιλήσω δανεικά, διότι είναι δανός και ο συντάξης νομοδότησης και θα με καταλάβει απευθεία. Ευχαριστώ λοιπόν, καλημέρα σας. Η σκιώδηση συγγήτρια μεταβαίνει στην Κίνα αυτή τη στιγμή με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κίνα και λυπάται πάρα πολύ που απουσιάζει σήμερα από την Επιτροπή μας. Είναι πραγματικά κρίμα και και το γεγονό ότι ταξιδεύει αυτή τη στιγμή. Θέλει να ευχαριστήσει τον ε, εισηγητή για τη γνωμοδότηση αυτή. Γενικά συμφωνεί, αλλά επίσης θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ε, είναι περισσότερη η ακρίβεια με την οποία αναφερόμαστε σε κάποια θέματα όπως είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας γιατί θεωρεί ότι στην Κίνα δεν τα χειρίζονται σωστά αυτά τα θέματα των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησίας. Είναι προβληματικό δηλαδή ένας Ευρωπαίος επιχειρηματίας να έχει στοιχεία ε, ε, και να μπορεί να επικοινωνεί με κινέζικες εταιρείες χρειαζόμαστε και πληροφορίες και ενημέρωση αξιόπιστη στην οποία μπορούμε να βασισόμαστε. Επίσης τα εμπορικά σήματα. Θεωρεί και ο δισηγήτρια ότι θα πρέπει να αναφέρονται στην νομοδότηση, καθώς επίσης και ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των προϊόντων των κινέζικων προκειμένου. Όπως λέτε και εσείς, γίνεται διάλογος αυτό το καιρό, αλλά ε, η σκιώδη συγγήτριά μας θέλει να ενισχυθεί ο διάλογος αυτό. Σας ευχαριστώ και προσβλέπει συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ας μιλήσω εγώ τότε, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ρούλε δεν είναι παρούσα. Εκπροσωπώ και την κυρία Μακράκιν. Νομίζω λοιπόν ότι η έμφαση που δίνει επιχειρηματή, ο εισηγητής στην επιτυχή ένταξη της Κίνας στο σύστημα του ΠΟΕ είναι σημαντική και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να κερδίσει στο παγκόσμιο επίπεδο από αυτό. Συμφωνώ με πολλές από τις κύριες συστάσεις της εκθέσεως, θα πρόσθετα και ορισμένες λίγο διαφορετικές αποχρώσεις. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό την προσπάθεια αυτή δημιουργίας, ε, ε, οικοδόμηση αυτή τη σχέση είναι και ένα τμήμα επικοδομητική κριτικής. Για παράδειγμα, για αντιμετώπιση θεμάτων διαφθορά. Μας έχετε δώσει μια πρώτη γεύση αυτού σχετικά με τι επενδύσει, αλλά πρέπει να μπει κάποιο στοιχείο ισορροπίας. και βεβαίω θέματα όπω η ασφάλεια των προϊόντων, που ξέρω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυρία Σάλντε Μόζε. Οι κεντρικέ αρχέ στην Κίνα γνωρίζουν πολύ καλά την ανάγκη εξασφάλιση τη ασφάλεια των προϊόντων. Αλλά η Κίνα είναι με τεράστια οικονομία και οι έλεγχοι που θεσπίζουν οι κεντρικέ αρχέ δεν φτάνουν μέχρι τι άκρε τη οικονομία αυτή. Χθε συζητήσαμε για φραγμού στο εμπόριο. Η κατάληξη σε συμφωνία ε, για μια συνολική ισορροπημένη προσέγγιση για μια προσέγγιση δηλαδή που να είναι βασισμένη σε στοιχεία για θέματα ασφάλειας των προϊόντων. Λέτε εδώ ότι η Κίνα εναρμονίζει τις εθνικές, τα εθνικά της πρότυπα με τα διεθνή πρότυπα. Θα πρέπει η Κίνα να μπει μέσα στην συζήτηση για την θέσπιση των διεθνών προτύπων, αυτό θέλω να πω εγώ και η χρήση των διεθνών προτύπων τους δίνει και ένα de facto πλεονέκτημα. Για παράδειγμα για τα αυτοκίνητα δεν έχουν πρότυπα για τις εκπομπές των ε, ε, καυσαερίων. Κάτι το οποίο αποτελεί φραγμό για αυτούς. Υπάρχει εδώ μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μέρος της συνολικότερης σχέσης. Και μου φαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ πιο επικοδομητικό παρά να επικρίνουμε μόνο το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στις εμπορικές συναλλαγές. Υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας διότι πρόκειται για μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και ξεκινώντας από πολύ διαφορετική βάση από την ευρωπαϊκή. Όταν θα μπει ωστόσο στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Για το IPR συμφωνώ με την κυρία Σαντεμόζε ότι οι ίδιοι οι Κινέζοι και οι κινέζικες εταιρείες εκμεταλλεύονται την προστασία που προσφέρει το IPR, έστω και διστακτικά. Προστασία δηλαδή των ε, ευρεσιτεχνιών. Υπάρχει μια κινέζικη εταιρεία η οποία έχει ε, υποβάλει τι περισσότερες ευρεσιτεχνίε μέσα σε ένα χρόνο από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο. Γνωρίζουν λοιπόν την αξία του συστήματος. Για να επιτύχει αυτή η ένταξη της Κίνας στο σύστημα του ΠΑΕ θα χρειαστεί και ενθάρρυνση των επιστημονικών και εμπορικών συναλλαγών ε, πολιτιστικών συναλλαγών και ούτω καθεξής. Μια ενίσχυση της πολιτικής αυτής. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα πούμε εδώ επίσης. Και αυτό κάνει και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου νομίζω. Πολύ ευχαριστώ λοιπόν θα συνεργαστούμε μαζί σας και ξέρω ότι η κυρία Μακλάρκιν θα καταθέσει και τροπολογίες λίγο πολύ, λίγο πολύ πάνω στι γραμμέ που σα εξήγησα. Η κυρία Ιβάνοβα, ε, ο κύριος Τενταφυλλίδης πρώτος ή εσείς πρώτοι. Κύριε Τενταφυλλίδη παρακαλώ. Ο κύριος Ντεγιόγκ είναι σκιώδη ηγητής για την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ ωστόσο τον εισηγητή. Ο κύριος De ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και ιδίω για τα όσα είπατε εσείς για την προστασία των διεθνών, ε, διεθνή προστασία μάλλον των ε, ε, δικαιωμάτων βιομηχανικής διοκτησίας. Η κυρία Ιβάνοβα παρακαλώ τώρα. Θα σας τα πω στα βουλγαρικά αυτή τη φορά. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι σκιώδη συγγήτρια για το θέμα αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και για μένα ως αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κίνα. Μπορώ να σας πω ότι συζητούμε ενεργά την έλλειψη ισορροπίας στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ευχαριστώ τον συνάδελφό μου, κύριο Λόκεγκορ, για τις θαυμάσιες προτάσεις που έχει καταθέσει. στο σχέδιό του και θα ήθελα να τονίσω δύο πτυχές που ίσως ήδη να τις έχετε θίξει, αλλά εγώ ήρθα με κάποια καθυστέρηση. Η πρώτη λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και εννοώ την συναλλαγματική ισοτιμία του Ιουάν, του κινέζικου νομίσματος. Δεν είναι βέβαια το κυριότερο πρόβλημα, ωστόσο είναι ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την έλλειψη αυτής της ισορροπίας στο εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Και το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που αναφέρθηκε ήδη αλλά ίσως πρέπει να συζητηθεί περισσότερο είναι το πρόβλημα του προστατευτισμού. Θα ήταν επικίνδυνο και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε μέτρα προστατευτισμού γιατί κάτι τέτοιο θα εντείνει τα προβλήματα αντί να τα λύσει. Είναι σημαντικό για μας να ακολουθήσουμε μια θετική γραμμή και αυτή τη θετική γραμμή ακολουθούμε άλλωστε στην αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Κίνα. Η θετική γραμμή είναι ανάγλυφη πραγματικά σε τούτην εδώ την έκθεση και γι' αυτό συγχαίρω τον εισηγητή. Πρώτα σας ευχαριστώ. Η κυρία Στάιλερ. Ίσως και άλλα μέλη. Έχουμε άφθονο χρόνο αν θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει ισορροπημένο ή όχι εμπόριο. Και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη την, τον οικονομικό πλούτο της Κίνας που όλο ένα και αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων και αγωθών. Θα πρέπει να προωθήσουμε έναν διάλογο με τις κινέζικες αρχές και αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε και για την αγορά εργασίας στην Κίνα. Να το δούμε με τις επιχειρήσεις μας, γιατί κανένας δεν έθιξε αυτό το ζήτημα. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε είναι κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας και να δούμε κατά πόσο στο μέλλον θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτό το διάλογο και τις συζητήσεις εν γέννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Στάιλερ. Υπάρχουν άλλα μέλη που θα ήθελαν το λόγο. Ο κύριος Νίλς Γιούκερ ε, Γιάκοψεν θα ήθελε να σχολιάσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα, θα θέλετε να μας δώσετε μία πρόγευση ή κάτι να μας πείτε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε σχόλιο ε, πρόσδεκτο. Α, όχι, είσαστε παρατηρητής. Καλώς. Ε, ο κύριος Λούκεγκαρτ έφυγε, ο κύριος ε, Κρόιτσμαλ συνομιλεί θερμά με τον γείτονά του. Κύριε Κρόιτσμαλ. Δεν ε, έχω πολλά να πω. Ε, θα... Έχω σημειώσει αυτά που είπατε. Θα τα διαβιβάσω στον κύριο Λούκεγκάρτ και αυτά θα ήθελα να πω προς το παρόν. Το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σημαντικό. Το θέμα του προστατευτισμού, της ασφάλειας των προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται για κάτι το καινούριο. θα δούμε και το θέμα των εξαγωγών τους, θα προβάλλουμε ένα προστατευτικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο προστασίας και όλα θα τα διαβάσω στον κύριο Λούκεγκάρ. Όπως ξέρετε, το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία που θα γίνει στις 10. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να διακόψω μέχρι τις 10 παρα 5 έτσι ώστε να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες ακριβώς στις 10. Θα σας δω λοιπόν τότε. Και να σας υπενθυμίσω ότι μετά την ψηφοφορία έχουμε κάτι σημαντικό. Ε, γιατί θα έχουμε μια συζήτηση με, για την περιαγωγή με βάση τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω λοιπόν να παραμείνετε για αυτή τη συζήτηση και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ε, δύναμη των καταναλωτών και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα προωθήσουμε την πολιτική μας. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Σήμερα το πρωί θα σας δώσω στις 10. Ευχαριστώ. Uh, um, Κυρίες και κύριοι, θα σας παρακαλούσα να καθίσετε όλοι, γιατί θα ήθελα να αρχίσουμε ακριβώς στις 10 τις ε, ψηφοφορίες. Έχουμε δύο ρολόγια με διαφορετική ώρα βέβαια. Εγώ δουλεύω με το αριστερό. Καθίστε σας παρακαλώ για να ψηφίσουμε. Ε, να έχετε και τις κάρτες σας, είστε βέβαιοι. Παρακαλώ. ADR um, Καλώς. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά την έκθεση του κυρίου Ροσφό, εναλλακτική τρόπη επίλυση των διαφορών. που αρευρίσκεται και ο εισηγητής. Θα θέλατε να πείτε δύο λόγια πριν περάσουμε στη ψηφοφορία, κύριε εισηγητά. Ο κύριος Ζωσφο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σε μεγάλη φόρμα μετά τις διακοπές και στρωνόμαστε στη δουλειά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν στην έκθεση αυτή. Οι πολιτικές ομάδες, οι ηγητές, συνεργάτες, βοηθοί. Νομίζω ότι για την έκθεση αυτή κάναμε μια προσπάθεια ε, να βρεθεί συνένεση και τα καταφέραμε σε όλες σχεδόν τις τροπολογίες, όλες τις συμβαστικές πλην μίας. Χαίρομαι γι' αυτό και πολύ δε περισσότερο που ήταν δύσκολη περίοδος γιατί χρειάστηκε να δουλέψουμε γρήγορα ε, με διαδοχικές επιστροφές από διακοπές. Επίσης έχουμε πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία προθεσμία στις 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουν στη Νομική Επιτροπή και στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου ε, στη συνέχεια. Λοιπόν, δουλέψαμε και γρήγορα και σωστά. Όλα αυτά γιατί τα κάνουμε. Ε, στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα πρώτα απ' όλα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για το πεδίο ε, εφαρμογής αυτών των τρόπων επίλυσης διαφορών αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σαφέστατο μήνυμα και ε, περιμένουμε νομοθετικό κείμενο επ' αυτών των θεμάτων. Θα είδατε κι εσείς από τις τροπολογίες που κάναμε με το γραφείο μου ότι κάθε φορά προσπαθούμε να έχουμε ως αφετηρία της απόψεις των συναδέλφων και ο συμβιβασμός να μην είναι αναγκαστικός, δηλαδή ότι εμεί έχουμε αυτή τη γνώμη και να την ασπαστείτε και οι υπόλοιποι, λαμβάνουμε υπόψη τι τροπολογίε των υπολείπων, όλων των πολιτικών ομάδων. Νομίζω είναι υποδειγματική η εργασία αυτή, τουλάχιστον από τη δική μα ε, ομάδα εργασία και χαιρόμαστε πάρα πολύ για το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρο, σα ευχαριστώ και για την προσέγγισή σα. Ε, πραγματικά αφιλείτε και στις δικές σας προσπάθειες και στο ταλέντο σας ε, τους συμβιβασμούς. Λοιπόν, Μπορεί να χρειαστεί κάποιος έλεγχος στην πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Τροπολογία παριθμών 1 του εισηγητού. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Δατά. Εγκρίνεται. Ποιος ε, δίνει το σήμα στους σοσιαλιστές και δημοκράτες σήμερα, ποιος είναι WIP για να σας κοιτάω. Η Κρίστελ Σάλτε για να ξέρω πώς θα είναι οι συσχετισμοί αν χρειαστεί έλεγχος. Λοιπόν, η τροπολογία 11 του Λουί Γκρέχ. Ε, ψηφοφορία κατά τμήματα η χωριστή που έχει ζητήσει η ομάδα των φιλελευθέρων. Τη βλέπετε στον κατάλογο ψηφοφορία. Τμήμα πρώτο ψηφί υπέρ. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα Νομίζω ότι χρειάζεται εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει η επαλήθευση, παρακαλώ. Ένα έλεγχο να κάνουμε για να δούμε αν ψηφίζουμε σωστά ως προς τους αριθμούς. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 κατά 10 υπέρ. Η τροπολογία 64 του εισηγητή ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 του εισηγητή ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η Τροπολογία 4 υπέρ του εισηγητή κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία 6 του κυρίου Τριανταφυλλίδη και της κυρίας Σβένσον. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 5 του κυρίου Φόξ ψήφι π. Κατά. Απορρίπτεται. Η 8 έχει αποσυρθεί. Η 9. Σφάπ και Μέγερ. Μάγερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 10. Φόξ ψήφι π. Κατά. Άποχες. Περνάει. Εγκρίνεται. Η 11. Δεν χρειάζεται. Συμβαστική ένα Ψήφι υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. Συμβαστική δύο. Κατά τμήματα που έχουν στήσει οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Δεν θα σας τη διαβάσω, την έχετε στον κατάλογο ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Εγκρίνεται. Δύο. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 2. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 14 υπέρ, 18 κατά. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τις υπόλοιπες τροπολογίες που καλύπτονται από τη συμβιβαστική, έτσι δεν είναι. Όχι. Πρέπει να πάμε στη συμβαστική 3 τώρα. Μάλιστα, συμβαστική 3 ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 27. Γκρέχ και Βάιλερ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 27. Πέρασε. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Μπορείτε να κανονίσετε ποιος δεν θα ψηφίζει, παρακαλώ. Έχουμε ένα ΕΛΚ υπεράριθμο. Θα να ψηφίζουμε με τους σωστούς του ΕΛΚ τώρα. Αρχίζει και πάλι η ψηφοφορία με του σωστού ε, ρυθμού ανά πολιτική ομάδα. Τι ψηφίζουμε την 27 μάλιστα. Ξαναψηφίζουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι ε, ψηφίζουν σωστά από το ΕΛΚ. 10 υπέρ, 21 κατά. Συμβαστική 9. Ψηφί υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη 32 του κυρίου Γκρέκ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 32. Εγκρίνεται 19 υπέρ 17 κατά. Η παράγραφος 6. Η τροπολογία 34 του κυρίου ε, Χουάν Νόκ υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 33 καταπίπτει. Και θα προχωρήσουμε μέσω στην 39. Ε, Με προφορική τροπολογία την οποία βλέπετε στον κατάλογο, δεν θα τη διαβάσω, ε, χρειάζεται, 39 με την προφορική ψηφή υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Καταπίπτει 39 και ερχόμαστε στη 40. Τμήμα πρώτο, τη ψηφοφορία έχει ζητήσει η ομάδα των φιλελευθέρων. Χάντς Πέτερ Μάγερ και Ανδρέας Φαπ, τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά επίσης εγκρίνεται. Α, τρίτο τμήμα, δεν το είχα καταλάβει, νόμιζα ήταν δύο. Υπέρ, α, ζητάει διαγραφή. Αν ψηφίσετε υπέρ της ε, τροπολογίας αυτής του τρίτου τμήματος, σημαίνει διαγραφή της παραγράφου, υπέρ της διαγραφής κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 41. Υπέρ, είναι του κύριου Σφάμπη, τροπολογία κατά. Συγγνώμη να σας ξαναδώ, δεν κατάλαβα. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η τροπολογία 42, πάξας. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 54. Κοράτσα Μπίλτ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 56. Έχει ζητήθει ψηφοφορία κατά τμήματα από τον εισηγητή. Τμήμα πρώτο, Μάλλον θα χρειαστεί ηλεκτρονική ψηφοφορία γι' αυτό. 56, πρώτο τμήμα. Αρχίζει. Α, τώρα περσεύει ένας συντηρητικός. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μεγάλη πλειοψηφία. Υποθέτω ότι το δεύτερο τμήμα θα καταπέσει τώρα. Η τροπολογία 55, καμφά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται 20-15. 57 Μάιερ και Σφάπ. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και πάμε στις νέες παραγράφους. 61 του εισηγητή, τροπολογία, υπέρ κατά εγκρίνεται, η 24 κατά καταπίπτει. 63 του εισηγητού, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν κρίνεται με 21 ψήφους. Υπέρ 14 κατά. 62 καταπίπτει. 64 έχει αλλάξει θέση. 65 εισηγητή υπέρ. Α, όχι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Δεν κρίνεται. 6 εισηγητή. Αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται επίση. Οκ. Τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία 69. η 67 έχει αποσυρθεί. Της κυρίας Κόρατσα Μπίλτ. Ψήφι πέρας 69 κατά εγκρίνεται. 68 της κυρίας Βάιλερ, υπέρ. Κατά, επίσης εγκρίνεται. 70 του κυρίου Μάντερς, υπέρ. Κα... Κατά. Ζητώ συγγνώμη, εδώ θα χρειαστεί έλεγχος γιατί δεν κατάλαβα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 70. Πέρασε. Εγκρίνεται 18-16. Συμβιβαστική 11. Ψηφίπε. Κατά. Εγκρίνεται. 75 ε, Α, έχει καταπέσει γιατί απορρίφθηκε 65 μάλιστα. 76 θα την ψηφίσουμε. Το κύριο Πουπάκη. Ψηφίπε. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 7, ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Συμβαστική κατά επίσης εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο. Πέρας. Εγκρίνεται 32 ψήφους υπέρ, καμία κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια τον εισηγητή, τον κύριο Ροσφό. Uh, and, um, so we look forward to you Ελπίζουμε να προασπίσετε τη θέση μας στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, να την προβάλλετε όπως πρέπει. Τώρα προχωράμε στην ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για το μέλλον του ΦΠΑ. Η συντάκτρια κυρία Ιβάνοβα, θέλετε κάτι να μας πείτε πριν από την ψηφοφορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδης για την γρήγορη αντίδρασή τους και άκρος αποτελεσματική γιατί είχαμε πολύ λίγο χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τη Γραμματή για την εξαιρετική αυτή εργασία. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τώρα. Συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά. Περνά, εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Τώρα Προχωράμε στην πρόταση συμβασμού 2. Τροπολογία συμβασμού 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 12, τροπολογία 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 καμφά αρχίζει η ψηφοφορία επί της 13 υπέρ μάλλον με συγχωρείτε ηλεκτρονική ήταν, πέρας, εγκρίνεται με 18 υπέρ και 14 κατά, 25 καμφέ. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 25. Πέρας. Εγκρίνεται 22 έναντι 13, 15 Διόγκ. Υπέρ. Κατά. Σαφέστατα εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα περνάμε τώρα στην, ε, μάλλον στις 22 και 23 που είναι παρόμοιες, αποτελούν προστίκη υπέρ, κατά, απορρίπτονται σαφέστατα. Τροπολογία συμβασμού 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 μπουζό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27 μπουζό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 5. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 5 τροπολογία συμβασμού. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 έναντι 11. 31. Χουανόκ. Προσθήκη στην τροπολογία συμβασμού. Αρχίζει η ψυχοφορία επί της 31. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 αρίας υπέρ κατά εγκρίνεται 33 της συντάκτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 35 καμφά υπέρ μάλλον ε, υπέρ παρακαλώ κατά απορρίπτεται σαφώς 37 χονόκ υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία συμβάσμου 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 44 τώρα. Καλπέλς υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβάσμου 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 8 υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε, τα έχασα, λέει ο πρόεδρο. Τροπολογία συμβιβασμού 8. Εγκρίθηκε, ωραία. Άρα τώρα ψηφίζουμε την 55. 55. Με συγχωρείτε, κάπως τα είχα χάσει. 55 αρχίζει η ψηφοφορία. 55. Κορέια Campos Πέρας. Απορρίφθηκε. 56. Κάλο ετούν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν ψήφισαν και τόσο πολύ. Πέρασε με μία ψήφο μία επιπρόσθετη. 57 μπουσόι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58 Ντε Γιόγκ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Μάλλον ε, ηλεκτρονική, η οποία και αρχίζει για την 59. Πέρας. Απορρίφθηκε. 60 ταραμπέλα υπέρ. Α, με συγχωρείτε, ηλεκτρονική αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 60, πέρας. Απορρίφθηκε. 61 μπουσόι. Υπέρ. Κατά. Σαφέστατα εγκρίθηκε τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότηση στο σύνολο του ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία ως προς το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Πέρας. That's carried by 31... 31 ψήφοι υπέρ, κανείς κατά και 5 αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ιβάνοβο πιστεύω ότι θα προωθήσει το θέμα στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών. Όπως πρέπει. Τελική ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό. Ο κύριος Κουζουτσινίκ είναι εδώ. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια. Εάν υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία γιατί το θέμα αυτό του προϋπολογισμού απασχόλησε όλες τις επιτροπές. Ως προς τις τροπολογίες, στη δική μας επιτροπή τουλάχιστον, νομίζω ότι όλοι υποστήριξαν τη βασική ιδέα ότι θα πρέπει να ε, υπερασπιστούμε την εσωτερική μας αγορά. Είχα ορισμένες ε, αμφιβολίες για τις τροπολογίες Κρόιτσμαν, αλλά νομίζω ότι μπορώ να τις υποστηρίξω αφού το σκέφτηκα. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης έχουμε και εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και ίσως θα θελήσουν να σχολιάσουν καθώς τις διατρέχουμε. Uh, I see Stefan Asoro is certainly here, I think. Uh, I think if they'd like to signal when they, when they wish to make... Όποτε θέλετε το λόγο να μας το πείτε, να μας το λέτε εγκαίρως. Θα ψηφίσουμε καταρχήν την έκθεσή σας και διαφορετικά τις γραμμές του υπολογισμού, ξεχωριστά μάλλον. Ας δούμε την έκθεση καταρχήν και μετά ενδεχομένως και η Επιτροπή να θελήσει να παρέμβει στο τέλος της ψηφοφορίας ή ενδιάμεσα. Ένα σαλδεμόζε Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα οι δύο καταπίπτει. 2. Υπέρ. Περνά. 5. Κουν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τέσσερα Γκρέκ που είναι προσθήκη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έξι. Σαλτεμόζε. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 6. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 7. Πάξας. Με ξεχωριστή ψηφοφορία, όπως ζήτησαν οι φιλελεύθεροι, βλέπετε λοιπόν στα χαρτιά σας πως έχει ξεχωριστεί πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Το ψηφίζουμε τώρα. Μάλλον αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Επί του δευτέρου τμήματος της τροπολογίας αυτής, της 8. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9 με μια προφορική που βλέπετε στο κάτω μέρος του καταλόγου ψηφοφοριών από τον εισηγητή. Είναι η προφορική υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 και 11 που είναι παρόμοιες υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνονται. Άρα τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, ηλεκτρονικά. Το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία ενκρίθηκε Εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ, καμία κατά και τρεις αποχές. Τώρα θα δούμε τις γραμμές ξεχωριστά, την κάθε γραμμή ξεχωριστά του προϋπολογισμού. Θα σας, μπορούμε να τις δούμε unblock, μπορούμε να τις ε, ψηφίσουμε unblock ή πρέπει να δούμε γραμμή προς γραμμή να τις εκφωνήσω ξεχωριστά. Ναι, πρέπει να το κάνουμε αυτό για διαδικαστικούς λόγους. Θα τις δούμε αναγραμμή λοιπόν. Θα τις δούμε unblock και ενδεχομένως η Επιτροπή να θελήσει να σχολιάσει αφού ψηφίσουμε. Η Επιτροπή μπορούμε να παρέμβουμε πριν από την ψηφοφορία. Ναι, κυρία Βανχέβεν. Εξ ονόματος της Επιτροπής έχετε το λόγο. Ε, εκπροσωπώ τη συνάδελφο και είμαι υπεύθυνη για το Solvit. Όπως σας έλεγα, είμαστε υπεύθυνοι για το Solvit και το σύστημα της ενιαίας αγοράς και ετησίως μας ε, μιλάτε για μια σειρά γραμμών κονδυλίων. Από ό,τι κατάλαβα φτάναμε στο 1,2 και από ό,τι κατάλαβα, ο, ο εισηγητής ήθελε να αυξηθούν οι πιστώσεις, αλλά ε, δεν ξέρω κατά πόσο ε, έχει νόημα να μιλήσω τώρα για την γραμμή όσον αφορά το Solvit. Πρόκειται για την 7003. Λέει ο πρόεδρος προς τον εισηγητή. Τι θέλετε να πείτε. Θα ήθελα να πω, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη της δράσης μας, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Solvit, αλλά και για την Ευρώπη, η οποία ολοένα και επεκτείνεται. Μιλήσαμε για 1,3 εκατομμύρια πέρσι στις δεσμεύσεις υποχρεώσεων που θα δαπονηθούν μέχρι το τέλος του έτους. Άρα δεσμευόμαστε γι' αυτό. Για το μέλλον, για του χρόνου, επειδή διανύουμε τη δέκατη επέτειο του Solvit, θα προβούμε και σε άλλες δραστηριότητες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επεκτείνεται και η Ευρώπη. Γι' αυτό μιλάμε για προβλέψεις 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να περάσει ως προφορική τροπολογία. Έτσι τουλάχιστον είχαμε καταλάβει. Μπορώ να σας δώσω λεπτομεριακές επεξηγήσεις για το πώς φτάσαμε στο 1,4, αλλά αυτό ήθελα να σας πω καταρχήν. Θα το επιβεβαιώσει ο εισηγητής τι θα ήθελε ακριβώς να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο σε σχέση με το Solvit. Νομίζω ότι οι συζητήσεις σε αυτή την Επιτροπή ε, ήταν ιδιαίτερα ζωηρές. Οι συνάδελφοι με γνωρίζουν. Εγώ είμαι αρκετά μετριοπαθής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και όταν πρόκειται για τη συγκεκριμένη πρόταση, έλαβα υπόψη τη θέση των συναδέλφων που πρόωθησαν τη θέση των καταναλωτών. Λυπάμαι γιατί ακούσαμε αυτή την υπόδειξη τώρα κατά την ψηφοφορία τη στιγμή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε. Επομένως, προτείνεται να γίνει δεκτό το 1,4 εκατομμύρια που ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει την τελική απόφαση. Ναι βεβαίως. Σας ευχαριστούμε. Εγώ είμαι υπεύθυνο για το φόρουμ της ενιαίας αγοράς. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή ε, σας στην οργάνωση του φετινού φόρουμ. Είναι δύσκολο βέβαια, ε, κοντεύουμε τον Οκτώβριο τον Οκτώβριο που γίνεται δηλαδή. Μία μικρή δήλωση τώρα για του χρόνου. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ προτείνει για του χρόνου να, ε, οργανωθεί το, να διοργανωθεί το φόρουμ σε, ε, σε όλες τις χώρες μέλη σε, ταυτόχρονα την ίδια εβδομάδα για να εξηγήσει στους πολίτες περί τίνος πρόκειται και να προσθέσουμε την ε, περιγραφή σε αυτό εδώ του φόρουμ της έννοιας αγοράς. Μια μικρή λοιπόν διευκρίνηση. Έχετε μια τροπολογία σχετική, έτσι δεν είναι. Εμένα μου φαίνεται κάπως δυσάρεστο ότι η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, δεν ήρθε σε επαφή με τον εισηγητή πριν να καταθέσει τα θέματα, τα πράγματα αυτά. Εγώ υποστηρίζω τις, ε, εγώ τις υποστηρίζω τις ιδέες αυτές, αλλά γιατί τόσο καθυστερημένα. Γιατί υποβάλλονται τόσο καθυστερημένα. Πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Υποθέτω ότι έχει σχέση με τη χρονική διάρθρωση του προϋπολογισμού, το λεγόμενο timing. Και οι συγκητές ε, δούλεψαν σκληρά για να τα συνδιαθρώσουν όλα αυτά και βεβαίως όλα τα μέλη δεν ήταν παρόντα. Πάντως θα πάει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και θα επανέλθει σε εμά για το τελικό OK. Σημειώνουμε τα σχόλιά σας. Για το χρόνο θα πρέπει να εξετάσουμε το χρονοδιάγραμμα του προπολογισμού για να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε μια πληρέστερη συζήτηση. Προχωρούμε λοιπόν χωρίς βέβαια να έχουμε πλήρη γνώση. Έχουμε τώρα και άλλα κονδύλια και τις σχετικές αιτήσει. Τα ψηφίζουμε ξεχωριστά αυτά. Αν χρειαστούμε τις συμβουλές του εισηγητού θα μας τις δώσει. Τώρα λοιπόν, οι 7.000 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7.001 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7.002 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7003 μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρα εκπίπτει 7003 χωρίς την προφορική τροπολογία. 7004 εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία το κ. Κρόιτσμαν αν δεν κάνω λάθος. Θέλατε εσείς να μιλήσετε. Θέλω μόνο να πω ότι πρώτα θέλω να ευχαριστήσω την ΙΜΚΟ που επανέρχεται στα θέματα εποπτείας της αγοράς. Το ιστορικό σας είναι εξαιρετικό. Η ΔΕ Κομισιόν υποστηρίζει την προφορική τροπολογία του κ. Κρότσμαν διότι θεωρούμε ότι καθιστά την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος πολύ ευκολότερα εφικτή. Υποστηρίζουμε λοιπόν την τροπολογία του κ. Κρότσμαν. Αντιληφθήκατε όλοι περί τίνο πρόκειται, δηλαδή τι, είναι η τροπολογία Κρότσμαν. Κάνα λοιπόν. Και έχετε όλοι αντίγραφο. Άρα την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάνω σε 7.004 εκπίπτει. Εδώ λίγη η ψηφοφορία αυτή. Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν θέλουν να πούν κάτι για τον προπολογισμό. Όχι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόσουτσνικ που έκανε την συνέταξη, την πρώτη του έκθεση για τον προπολογισμό, για λογαριασμό μας και θα συζητήσουμε πλέον με την Επιτροπή Προπολογισμών. Και όσοι δεν θα παραμείνουν για την επόμενη πολύ σημαντική παρουσίαση για την περιαγωγή, ας ε, αποχωρήσουν ε, τις αιθούσει, όσοι δεν θα μείνουν δηλαδή. Σύντομη διακοπή δύο λεπτών. Ryman. So, ladies and gentlemen, can we um, Ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημαντικό θέμα στη μερική διάταξή μας, δηλαδή η έναρξη της εργασίας μας σε ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό θέμα που έχει βέβαια και μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και ενώ την προτινόμενη αναθεώρηση της ε, οδηγίας για την περιαγωγή και τα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Πολύ εξημών θα έχετε εργαστεί στα δύο προηγούμενα πακέτα περιαγωγής, όπου η παρούσα Επιτροπή είχε παίξει σημαντικό ρόλο μαζί με την, βιομηχανία, με την Επιτροπή Βιομηχανίας, για να, όπου θέσαμε δηλαδή τα θέματα των καταναλωτών. Αρχίζουμε τώρα τη δουλειά μας με την κυρία Κόρχολα, που είναι η συγγήτριά μας η Επιτροπή Βιομηχανίας ακόμη δεν έχει ορίσει εισηγητή, έτσι λοιπόν προηγούμαστε λίγο, αν και νομίζω ότι άκουσαν ε, χθες εκεί τα μέλη ε, την, ε, ε, την παρουσίαση που θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και εμείς σήμερα του κυρίου Τέραβα και που θα εξηγήσει την αξιολόγηση του αντικτύπου της ε, επανεξέτασης του κανονισμού περί περιαγωγής. Θα παρακαλέσω τον, τον κύριο Τέραβα να κάνει την παρουσίαση. Μετά θα παρακαλέσω την κυρία Κόχολα να κάνει ε, σχόλια. Δεν ξέρω αν έχουμε όλους τους και όλες των πολιτικών ομάδων. Νομίζω θα προβλέψουμε μία ώρα για το θέμα αυτό. Άρα θα παρακαλέσω την Κομισιόν, τον κύριο Τέραβα, να κάνει την ε, σχετική παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Ευχαρίστως βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω την πρότασή μας για την αναθεώρηση του κανονισμού περιαγωγής που καταθέσαμε ήδη από τις αρχές Ιουλίου, όπως είπατε. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω την αιτιολόγηση, όπως την βλέπουμε, της πρότασής μας και να φωτίσω τις επιπτώσεις που θεωρούμε ότι θα έχει η πρότασή μας στους τελικούς χρήστες της περιαγωγής. Πριν από μπω στις λεπτομέρειες, ας αρχίσω εξηγώντας το μέγεθος της ε, αγοράς περιαγωγής καθώς και τη μορφή του ανταγωνισμού. Όταν μιλούμε για την αγορά περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούμε για 5 δις ευρώ περίπου που είναι περίπου το 4% των συνολικών εσόδων από την κινητή τηλεφωνία. Και αν εξετάσουμε την ανάλυση των διαφόρων υπηρεσιών περιαγωγής θα δείτε ότι η φωνητική τηλεφωνία εξακολουθεί και είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εσόδων, 71% δηλαδή, εξακολουθεί να είναι η φωνή, δηλαδή τα τηλεφωνήματα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι οι υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων που φτάνει περίπου στα 20% αλλά αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα και η αγορά μεταφοράς δεδομένων γενικά είναι ε, σημαντική και θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια λόγω της αυξανόμενης σημασίας της. Σχετικά τώρα με την διαδικασία επανεξέτασης μέχρι τέλους του, Ιουνίου φέτος είχαμε την υποχρέωση να κάνουμε την επανεξέταση. Κάναμε λοιπόν διαβουλεύσεις αρχίσαμε τον προηγούμενο χρόνο στις αρχές, δηλαδή φτάσαμε μέχρι το Φεβρουάριο φέτος, έχουμε προτείνει ορισμένες επιλογές, κανονιστικές επιλογές και κάνουμε τώρα τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων. Και θα καταλήξουμε, καταλήξαμε μάλλον στη νέα πρόταση Ιουλίου, του Ιουλίου 2011. Αν εξετάσετε τώρα πιο προσεκτικά την ε, κατάσταση του ανταγωνισμού και την εξέλιξη του ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής, δηλαδή το τι επέφερε η εφαρμογή του κανονισμού μέχρι τώρα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, πρώτα θα δείτε ότι ο κανονισμός περιαγωγής και οι operators των, ε, της κινητής τηλεφωνίας συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του κανονισμού Μειώθηκαν επομένω οι τιμές, αυτό είναι καλό νέο για τους ε, καταναλωτές. Από την άλλη μεριά όμω, παρόλο που μειώθηκαν οι τιμέ. βρίσκονται λίγο πολύ ε, εκεί που προβλέπουν οι κανονισμοί, δηλαδή δεν έχουν μειωθεί πολύ περισσότερο. Ο ανταγωνισμός δεν είναι ακόμη αποτελεσματικός, σε αυτό συμφωνούν όλοι οι ε, συμμετέχοντες όλοι οι φορείς και εξακολουθούν και υπάρχουν οι σχετικές δυσχέρειες. Αν εξετάσετε τώρα τον πίνακα της εξέλιξης των τιμών, πρώτα για τη φωνητική τηλεφωνία και μετά για τα δεδομένα, στον πρώτο πίνακα για την τιμή των τηλεφωνημάτων, θα δείτε την κόκκινη διακεκομένη γραμμή που είναι οι κορυφές, τα ανώτατα δηλαδή όρια και οι νυν τιμές που βλέπετε ότι προσεγγίζουν πάρα πολύ ε, στα όσα προβλέπει ο κανονισμός, τα ρυθμιστικά ανώτατα όρια δηλαδή. Δεν έχουν μειωθεί πολύ περισσότερες οι τιμές. Θα δείτε τώρα, θα δείτε ότι δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός και επομένως οι οπερατέρ δεν έχουν μειώσει σημαντικά τις τιμές πέραν των όσων προβλέπονται από τον κανονισμό. Στον επόμενο πίνακα θα δείτε τα δεδομένα, δηλαδή την εξέλιξη των τιμών της μεταφοράς δεδομένων με διαφορετικά τρίμηνα, ξεκινώντας από το τέλος του 2007, για, πρώτο, για κάθε τρίμηνο μάλλον, οι δύο πρώτες στήλες, ίσως δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, θα σας το εξηγήσω, οι δύο πρώτες στήλε είναι οι λιανικές τιμές του τελικού χρήστη. Ενώ το πορτοκαλί και το πράσινο είναι οι χονδρικές, οι τιμές χονδρικής δηλαδή μεταξύ επομένως ε, ε, των οπερατέρ. Και αυτές έχουν μειωθεί περισσότερο. Το, το ρυθμισμένο κενό τώρα είναι στα 50 cent του ευρώ. Στα 50 λεπτά του ευρώ δηλαδή. δηλαδή. Αλλά βρίσκονται περίπου μετά τον ανταγωνισμό στα 40 λεπτά. Ταυτόχρονα, κατά μέσον όρο, ο καταναλωτής πληρώνει παραπάνω από ένα ευρώ για κάθε megabyte περιαγωγής δεδομένων και ακόμη υψηλότερες τιμές για off-net data sessions, εκτός δικτύου δηλαδή. Επομένως έχει αυξηθεί το περιθώριο. Άρα οι ε, πάροχοι των υπηρεσιών αυτών ε, αποκομίζουν πολύ σημαντικά κέρδη. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπει κανείς ποιο είναι το κόστος της παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής. Και αυτά είναι στοιχεία του Μπέρεκ που συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα ανά και έχουν ε, πολύ αξιόπιστα δεδομένα και οι οποίοι υπολογίζουν πέραν των τιμών έχουν υπολογίσει και την δομή των ε, κλήσεων που δείχνει ότι για κλήσεις περιαγωγής το πραγματικό κόστος παροχής ενός λεπτού είναι μεταξύ 5 και 8 λεπτών του ευρώ. <clears throat> για τα μηνύματα SMS είναι μεταξύ 1,5 και 2 λεπτών. Για τα δεδομένα το κόστος είναι μεταξύ 8,5 και 12 λεπτά του ευρώ ανά μεγαμπάιτ. Βλέπετε λοιπόν τα τεράστια περιθώρια που διαθέτουν αυτή τη στιγμή για την αποκομιδή κέρδους η, η παρόχη των υπηρεσιών αυτών. Αν εξετάσετε τώρα ποια είναι τα βασικότερα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες στρατηγικά, στρατηγική φραγμή, κανονιστική και διαρθρωτική. Μας ζητήθηκε να εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες της αγοράς περιαγωγής και τα σφάλματά της που αυτά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και στο επίπεδο της χοντρικής και στο επίπεδο της λιανικής. Στο επίπεδο της λιανικής στο επίπεδο του καταναλωτή δηλαδή, δεν υπάρχει σημαντική επιλογή σε ό,τι αφορά την χρήση υπηρεσιών περιαγωγής, διότι η περιαγωγή δεν αποτελεί παρά μόνο ένα τμήμα ε, μιας, ενός συνολικότερου πακέτου κινητής ε, τηλεφωνίας. Υπάρχει και μια έλλειψη διαφάνειας, η αναζήτηση είναι και χρονοβόρα, είναι γνωστό αυτό, και τα τιμολόγια της περιαγωγής δεν είναι παρά ένα τμήμα μόνο μια, ενός μακρού καταλόγου τιμών. Είναι δύσκολο λοιπόν για τον καταναλωτή να βρει ακριβώς ποιες είναι οι τιμές της περιαγωγής που θα χρεωθεί τελικά. Πιστεύουμε ωστόσο ότι αυτό μπορεί να αλλάξει εάν οι υπηρεσίες περιαγωγής μπορούν να αγοράζονται ξεχωριστά από το υπόλοιπο πακέτο ε, υπηρεσιών τηλεφωνικής, ε, συγνώμη, ε, ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τώρα στο επίπεδο των ε, παρόχων. Ο αποκλισμός των, των εικονικών υπηρεσιών οδηγεί στην δυσκολία να εντάσσονται νέοι πάροχοι διότι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν ευθέω με αλλοδαπούς παρόχους, άρα χρειάζεται να αγοράζουν τις, τις υπηρεσίες περιαγωγής από, τον, ε, ε, από την εγχώρια αγορά, που συνήθως βρίσκονται άνω του ρυθμισμένου ορίου. Είναι δύσκολο λοιπόν να υπάρξει ανταγωνισμός. Και τέλος, η κατάσταση του ανταγωνισμού επιβαρύνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, πραγματική εναλλακτική επιλογή, υποκατάστατο των υπηρεσιών περιαγωγής. Υπάρχουν όμως κάποιες δυνατότητες. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το δίκτυο Wi-Fi ή IP ή να αγοράσει κανείς μια κάρτα κινητής τηλεφωνίας στην χώρα όπου επισκέπτεται. Αυτά όμως δυσχεραίνουν την ε, κατάσταση γιατί η περιαγωγή υποτίθεται ότι είναι ε, κάτι το εύχριστο. Επομένως ο καταναλωτής εάν θέλει να βρει άλλες εναλλακτικέ επιλογές πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια. Επομένως οι εναλλακτικέ αυτές επιλογές δεν έχουν ασκήσει ανταγωνιστική πίεση στους ε, παρόχους κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών περιαγωγής. Είναι περισσότερο συμπληρωματικός ο χαρακτήρας τους. Καλώ. Ε, κάνει καλό συμπλήρωμα, αλλά δεν έχουν αλλάξει την δυναμική του ανταγωνισμού στην αγορά. Στην βάση αυτών έχουμε προτείνει, έχουμε καταθέσει μια πρόταση που θεωρούμε ότι είναι υπέρ του ανταγωνισμού και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα διαφορετικά προβλήματα που ανέπτυξα. Πρόκειται για μια διπλή προσέγγιση. Αφενός εισάγουμε έναν αριθμό διαρθρωτικών στοιχείων, δομικών στοιχείων, που δίνουν περισσότερες επιλογές στον καταναλωτή για υπηρεσίες περιαγωγής και δίνουν τη δυνατότητα νέων εισόδων σε περισσότερους ανταγωνιστές να μπουν δηλαδή στην αγορά περιαγωγής. Ταυτόχρονα προτείνουμε να συνεχιστούν, ε, να συνεχιστεί η εφαρμογή οροφών στις τιμές μέχρι ότου ε, υλοποιηθούν ε, τα διαφθορτικά μέτρα και καταλήξουν σε μείωση τιμών λόγω ανταγωνισμού. Να συνεχιστούν λοιπόν αυτές οι οροφές τιμών ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον του καταναλωτού και ως νέο στοιχείο σε σχέση δηλαδή με τον ισχύοντα κανονισμό, προτείνουμε να εισαχθούν αυτά τα safeguard price caps και για τις ε, ε, υπηρεσίες περιαγωγής. Έχει πολύ ακόμα. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε εν λεπτομερία τα ε, δομικά μέτρα, τα διαρθρωτικά μέτρα, για να δούμε πώς αυτά τα μέτρα μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική της αγοράς, θα ήθελα να πω ότι καταρχήν θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η αγορά είναι ανοιχτή σε πολλούς παρόχους, δηλαδή να μπορούν οι οικονομικοί φορείς πάροχοι να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Και υπ' αυτή την έννοια η πάροχη δικτύου στην αγορά σύμφωνα με την πρότασή μας, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε εναλλακτικούς παρόχους με βάση τις ε, ρυθμισμένες τιμές χονδρικής, έτσι ώστε να μπορούν εναλλακτικά πάροχοι να παρέχουν υπηρεσίες σε περιαγωγές. Από πλευράς καταναλωτών, από πλευράς ζήτησης, θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες επιλογές. Και αυτό μπορεί να γίνει αν επιτρέψουμε στους καταναλωτές να μπορούν να ε, αγοράζουν την περιαγωγή σε μια ξεχωριστή καθαρά υπηρεσία. Τώρα, επανερχόμενος την πρόσβαση χονδρικής, χονδρικών υπηρεσιών, υπηρεσιών χονδρικής και υποχρεώσεων, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα διπλό ευεργέτημα. Δηλαδή μπορούμε να ε, δούμε κατά πόσο μπορεί να μπει κανείς στην αγορά περιαγωγής και όποιος μπορεί να το κάνει, μπορεί να φτάσει σε ρυθμισμένες ε, ε, υποχρεώσεις και συμβάσεις στη χώρα, στην επισκεπτόμενη χώρα ή τα επισκεπτόμενα δίκτυα και από την άλλη πλευρά μπορεί να φτάσει σε μια συμφωνία με τον πάροχο από τη χώρα προέλευσης που είναι και η ευκολότερη λύση ιδιαίτερα για τους ε, μικρούς ας το πούμε καταναλωτές και έτσι θα μπορούσαμε να, έχουμε, να φτάσουμε σε ένα πανευρωπαϊκό ε, προσέγγισης. Τώρα σε σχέση, μιλήσαμε για τη χονδρική. Το δεύτερο θέμα είναι η αποδέσμευση, δηλαδή η χωριστή χρέωση των υπηρεσιών περιαγωγής. Η αποδέσμευση. Αυτό το χρειαζόμαστε διότι η πρόσβαση χονδρικής θα σήμαινε ότι μπορεί κανείς πολύ δύσκολα να ε, μπει στην αγορά. και ε, αν ένας πάροχος δεν είναι ακόμα παρόν στην εγχώρια αγορά, εάν υπάρχει το σκέλος της περιαγωγής, ε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κινηθεί. Άμα όμως υπάρχει αποδέσμευση, μπορεί κανείς να μπει στην αγορά. Μπορεί να μπει δηλαδή μόνο ε, αν αγοράσει μία κάρτα SIM χωριστή κάρτα SIM. Και αυτό βεβαίως επιβαρύνει την κατάσταση. Αν πρέπει να αλλάξετε SIM για να καλέσετε στο σπίτι σας, στο σπίτι σας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται το unbundling, η χωριστή χρέωση δηλαδή, η αποδέσμευση. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στις υπηρεσίες περιαγωγής Εάν δεν ήταν τόσο ευαισθητοποιημένοι ως προς την τιμολόγηση, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να μπει κανεί στην αγορά, ιδιαίτερα άμα θα ήθελε να μπορεί να συγκρίνει τις τιμές. Αν δούμε τα πρόσφατα στοιχεία, βλέπουμε ότι οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στην τιμολόγηση της παροχής υπηρεσιών στον τομέα της περιαγωγής. Αν μπορούμε δηλαδή να μπούμε στην αγορά με αυτές τις προσφορές μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει τις τιμές και να επιλέξει τον πάροχο που τον βολεύει, δηλαδή που είναι πιο δελεαστικός, που προσφέρει χαμηλότερη τιμή. Άρα αν μπορούν να αλλάξουν οι καταναλωτές, αυτό ασκεί πίεση και στους παρόχους. Πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Άρα ε, υπάρχει ενδιαφέρουσα ε, τιμολόγηση και από πλευράς των ε, παρόχων που προϋπάρχουν θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Ως προς το unbundling, την αποδέσμευση ή τη χωριστή τιμολόγηση θα πρέπει να είναι φιλική προς τον καταναλωτή. Θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης να αλλάξει από τον υπάρχοντα πάροχο σε έναν άλλο πάροχο για την περιαγωγή και θα πρέπει και οι εμπλεκόμενοι φορείς να προβάλλουν διαφάνεια για τον ε, καταναλωτή, ο οποίος να ξέρει ποιες είναι και οι εναλλακτικέ. Εμείς έχουμε προβάλει μία τεχνική λύση, τεχνική υφής, είναι βεβαίως ε, επικουρική, προαιρετική. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι προώθησης της αποδέσμευσης, του ε, unbundling σε αυτή τη διτή προσέγγιση, ο καταναλωτής με την ίδια κάρτα SIM έχει δύο παρόχους, μία για τις εγχώριες υπηρεσίες και έναν εναλλακτικό πάροχο για την περιαγωγή. Άρα δεν χρειάζεται να αλλάξει κάρτα SIM και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ένα εύχριστο σύστημα, ιδιαίτερα φιλικό για τον καταναλωτή, για τον πελάτη. Όπως ήδη προείπα, Μαζί με τα διαρθρωτικά μέτρα θα πρέπει να έχουμε και τιμολογήσεις, ανώτατα όρια τιμολογήσεων, πριν τεθούν σε πλήρη εφαρμογή τα διαρθρωτικά μέτρα. Θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους οικονομικούς φορείς και η προστασία του καταναλωτή. Στην πρότασή μας επίσης προβλέπουμε ότι θα υπάρχει υπάρχουν ανώτατα όρια λιανικής μέχρι το 2016 περιλαμβάνοντας ε, και τα, την τιμολόγηση, τη λιανική τιμολόγηση περιαγωγής, διότι μέχρι το 2016 τα διαρθρωτικά μέτρα θα τεθούν πλήρως σε εφαρμογή. Ως προς το unbundling, τη χωριστή χρέωση, όπως σας είπα, Δίνουμε στους ε, οικονομικούς φορείς δύο χρόνια έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα τουλάχιστον μέχρι το 2014. Και στη συνέχεια θα ε, φτάσουμε στα τελικά ευεργετήματα προς τον καταναλωτή. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, εάν υπάρχει μία λύση, μία ανταγωνιστική λύση, για τους ε, καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι θα μπορέσουν να προβάλλουν εναλλακτικές τιμές, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Να υπάρχουν δηλαδή ανταγωνιστικές συναλλαγές πριν τεθούν σε εφαρμογή καθαρά τεχνικές λύσεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένουμε μέχρι το 2014 ε, για να ακολουθήσουν φθήνουσα πορεία οι τιμές, οι τιμολογήσεις. Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι μέχρι το 2016 η αγορά θα έχει προσαρμοστεί πλήρως. Μέσα στα πλαίσια αυτής της δυναμικής. Εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει πλήρης αναθεώρηση του κανονισμού περί περιαγωγής το 2015 και υπ' αυτή την έννοια θα μπορέσουμε να αποτιμήσουμε όλα τα στοιχεία του κανονισμού. Άρα υπάρχει αυτή η διασφάλιση, δηλαδή αν ε, δεν ε, προχωρήσουν τα πράγματα όπως προβλέπουμε, θα αποτιμήσουμε την κατάσταση εκ νέου το 2015. Ως προς την, ε, τη μελέτη αντικτύπου, εμείς την αναθεώρηση αυτή σκιαγραφίσαμε και προβάλαμε συγκεκριμένες εναλλακτικές για τον αναθεωρημένο κανονισμό. Θεωρούμε, αποτιμήσαμε τα στοιχεία υποποιωτικούς όρους και φτάσαμε σε λίγες εναλλακτικές λύσεις, σε ένα περιορισμένο κατάλογο, όπου έγινε ένας εις βάθος οικονομικός απολογισμός για να δούμε ποιες είναι και, ποιος είναι και ο αντίκτυπος στους καταναλωτές. Επίσης είδαμε ποιο είναι το κόστος εφαρμογής από την άλλη πλευρά. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αυτές τις λίγες εναλλακτικές. Έχουμε την τρέχουσα προσέγγιση θα μιλήσουμε για διαφάνεια και μέτρα χονδρικής, καθώς και τις χρεώσεις roaming από την πλευρά λιανικής. Άρα είχαμε ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών λύσεων που μετά από την ε, προκαταρκτική ανάλυση μας οδήγησε σε έναν ε, βραχή κατάλογο, περιορισμένο κατάλογο εναλλακτικών, δηλαδή θα συνεχίσουμε με την ε, τρέχουσα προσέγγιση των ανώτατων τιμών τιμολόγησης γιατί εδώ θα πρέπει να δούμε τις διάφορες εναλλακτικές. Η τρέχουσα προσέγγιση λοιπόν είναι η καλύτερη από όσο μπορούμε να κρίνουμε. Η δεύτερη εναλλακτική είναι η χαμηλότερη προσέγγιση ως προς τις ε, τιμολογήσεις και αυτό σημαίνει ότι θα ρυθμίσουμε τις ε, τιμές ε, λιανικής, οι οποίες θα προσεγγίζουν τις τιμές ε, χονδρικής για να αποτιμήσουμε το κόστος περιαγωγής. Και η τρίτη εναλλακτική είναι ο συνδυασμός των διαρθρωτικών μέτρων και των τιμολογήσεων ρύθμισης και διασφάλισης. Εάν δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις εναλλακτικές, και την ποιοτική την ποιοτική τους προσέγγιση βλέπουμε ότι δεν μεταφέρουμε τις μειώσεις της χονδρικής στη λιανική και έτσι η, η εικονική παροχή δεν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν ε, στην αγορά διότι υπήρχε διαφορά χάσμα μεταξύ χονδρικής και λιανικής. Επίσης, ως προς τις ανώτατες τιμολογήσεις, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλές υπηρεσίες για όλους τους χρήστες και έτσι είναι πολύ δελαστική αυτή η προσέγγιση. Όμως αυτά τα ευεργετήματα είναι περιορισμένα χρονικά. Δεν θα αντιμετωπίσουμε τα καθαρά διαρθρωτικά μέτρα και δεν θα βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό. Τέλος, ως προς τα ε, διαρθρωτικά μέτρα και τις ε, τιμολογήσεις διασφάλισης, θεωρούμε ότι θα έχουν επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και θα υπάρχει δυνατότητα νέων, θα υπάρχουν νέες δυνατότητες ανταγωνισμού. Ο καταναλωτής θα έχει διάφορες εναλλακτικές λύσεις και έτσι θα προβάλλουμε μία βιώσιμη λύση χωρίς να χρειάζεται μία μακροχρόνια τιμολόγηση ως προς την εκτίμηση της, ε, των οικονομικών αντικτύπων βλέπετε τα ευεργετήματα εδώ, τους αντικτύπους, σε σχέση με την ε, ανώτατη τιμολόγηση βλέπουμε ότι ο καταναλωτής θα έχει ένα μεγάλο ευεργέτημα. Αυτό το κρίνουμε για την περίοδο 2012 μέχρι 2014, 1,4 δις ευρώ, συγκρίνοντας ε, με το βασικό σενάριο της τρέχουσας προσέγγισης. Η διαρθρωτική λύση και οι τιμολογήσεις ε, διασφάλισης μας οδηγούν σε μία σταθερότητα. Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά ως προς την ε, προσέγγιση της τιμολόγησης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η, βασική μας προσέγγιση αφορά την ανώτατη τιμολόγηση ε, διασφάλισης. Και αυτό μέχρι το 2014. Μιλάμε για 1,2 δις. Πρόκειται για έναν συντηρητικό υπολογισμό. Ο πραγματικός αντίκτυπος θα είναι πιο ευεργετικός για τον χρήστη μέχρι τότε. Από την άλλη πλευρά τα στοιχεία αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος εφαρμογής που είναι πολύ σημαντικό. Κρίνουμε ότι για την τεχνική λύση που προαναφέραμε, την δυτή αυτή προσέγγιση, κρίναμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται από τα στοιχεία του φορέα αυτού, δηλαδή μιλάμε για 300 εκατομμύρια σε επίπεδο βιομηχανίας, δηλαδή κάτω από 10% των ετησίων εσόδων από την περιαγωγή ή 0,2% του ετήσιου, των ετήσιων εσόδων. Και τη στιγμή που θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα από την από πλευράς τιμολόγησης βλέπουμε ότι θα πρέπει καταρχήν να προϋπάρξουν επενδύσεις για να φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα. Επενδύσεις από τους παρόχους δηλαδή. Άρα η διαρθρωτική λύση μας οδηγεί σε μία μακροχρόνια λύση. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι αυτό αποτελεί μία επένδυση που αξίζει τον κόπολο να γίνει. Αυτή είναι μία από τις ενδεχόμενες τεχνικές λύσεις. Εάν υπάρχουν λιγότερο δαπανηρές λύσεις θα τις εξετάσουμε. Αλλά θα πρέπει οι εναλλακτικές, εάν υφίστανται, να οδηγήσουν στο ίδιο ευεργέτημα έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών. Τέλος, η συνολική αποτίμηση μας ε, ε, οδηγεί στα διαρθρωτικά μέτρα έναντι των ανώτατων τιμολογήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος, υψηλότερος ανταγωνισμός, περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή και μακροχρόνιες επιπτώσεις στον τομέα των ρυθμίσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, με χαρά να σας απαντήσω. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσίαση αυτή. Ε, η πρόταση είναι πολύ πιο περίπλοκη από την προηγούμενη βέβαια από κάποια έννοια. Αυτά τα θέματα της ανώτατης τιμής και της μείωσης των περιθωρίων των εταιριών ε, κινητής τηλεφωνίας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι αρκετά μεγάλο το περιθώριο μεταξύ των τιμών λιανικής και χονδρικής. Ε, είναι στοιχεία ενδιαφέροντα. Βεβαίω και για τις λύσεις, ε, κατά πόσο είναι διαρθρωτικές ή όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμά δεν είναι αυτό, είναι, είναι θέμα της Επιτροπής Μηχανίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, η σκοπιά του καταναλωτή, να μειώνεται το κόστος και ο χρόνος και ε, ε, λοιπά. Ε, θα παρακαλέσω τώρα τη συγγήτρια την κυρία Κόρχολα να ρίξει συζήτηση και έχουν ζητήσει και άλλοι συνάδελφοι το λόγο, κυρία Σάλτε Μόζε ε, και εγώ και κάποιοι άλλοι. Ο καθηγητής Κορέτα Κάμπος και εγώ βεβαίω ότι έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα στο παρελθόν ως και συγητή, αλλά ας αρχίσουμε από την συγγητρία μας, κυρία Κόρχολα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Όπως είπε στην αρχή ο Μάλκο, έχουμε αποκλειστικές ε, αρμοδιότητες εμείς στην Επιτροπή μας, αλλά και Επιτροπή Βιομηχανίας και θα πρέπει να δούμε και τα θέματα ε, των ε, τιμολογήσεων, ε, το timing του χρονισμού, των ε, τιμών λιανικής και ο καθένας έχει τη δική του αρμοδιότητα και θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό τον ε, επιμερισμό εργασίας. Η άλλη επιτροπή όμως από ό,τι άκουσα δεν έχει αρίσει ακόμα εισηγητή. Είναι το πρώτο πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος και από τη διαδικασία αυτή φάνηκε από την αρχή ότι αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς η κινητή τηλεφωνία. Όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν τα λεγόμενα ευφύ τηλέφωνα, smartphones και ε, πολύ περισσότερο χρησιμοποιείται το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. Οι σημερινές τιμές και τα τέλη είναι ε, πραγματικά υπερβολικά. Έχω ακούσει ε, για πολίτες που έχουν πάει διακοπές ε, σε άλλες χώρες και τους έχει έρθει ο λογαριασμός πάνω από 1000 ευρώ σε χώρες της Ένωσης επειδή ξέχασαν να κλείσουν το διαδίκτυο. Επίσης είναι πολύ εκπρόσδεκτη η πρόταση για ανώτατη τιμή στην περιαγωγή για τα στοιχεία για ε, το διαδίκτυο είναι ε, καλά μέτρα αυτά για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Είμαι ε, βέβαια ότι θα έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου για το ποια είναι τα καλύτερα μέτρα ε, από πλευράς ανταγωνισμού και βεβαίως θα έχουν τελικά και τη φυσική τους επίδραση στη μείωση των τιμών με μεγάλο ενδιαφέρον θα εργαστώ σε αυτό το θέμα και περιμένω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλια λοιπόν από άλλα μέλη της Επιτροπής, η κυρία Σαλντεμόζα. Ευχαριστώ. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ακόμα δεν έχει ορίσει σκιώδη συγητή. Μιλώ εξ ονόματο του εαυτού μου προ το παρόν, προσωπικά τελείω. Ε, σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σα και έχει σημασία όντω να κάνουμε κάτι ε, και να αντιμετωπίσουμε και τα διαρθρωτικά προβλήματα των αγορών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα. Πλην όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον τελικό χρήστη, τον καταναλωτή. Όπως είπε και η κυρία Κόρχολα, παίρνουμε όλοι πολλά email από συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, που είναι πάρα πολύ ε, λυπημένοι από το λογαριασμό τη λυπητερή που τους έρχεται μετά τις διακοπές σε άλλες χώρες. Εμείς δεν μπορούμε να ζητάμε από τους καταναλωτές ε, να κάνουν διάφορες επιλογές. Δεν θα το κάνουν. Οι περισσότεροι ταξιδεύουν μια φορά το χρόνο ή δύο φορές στο εξωτερικό. Τι σκέφτονται τώρα να πάνε να βρουν άλλη κάρτα SIM, να δουν ποια άλλη εταιρεία κάνει ποια περιαγωγή. Είναι ανεδαφικά αυτά, δεν είναι ρεαλιστικά. Εμείς που ταξιδεύουμε τόσο πολύ και είμαστε τόσο συνηθισμένοι να πηγαινοχόμαστε στο εξωτερικό, ε, μπορεί να το σκεφτόμαστε αυτό, αλλά πολλοί καταναλωτές δεν το πράττουν. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για τις ανάγκες της αγοράς και τις διαρθρωτικέ αλλαγές, αλλά να ε, βεβαιωθούμε ότι οι καταναλωτές δεν θα ε, παραγωνιστούν ή δεν θα υποχρεωθούν να κάνουν πάρα πολλές επιλογές θα πρέπει και στον καταναλωτή να υπάρχει ανώτατη τιμή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, δεν είναι εναλλακτικά μεταξύ τους αυτά. Θα κάνουμε και τι διορθωτικέ αλλαγές, αλλά και την ανώτατη τιμή στη λιανική. Και όχι εικονική οροφή, πραγματική οροφή, όχι μόνο στις τιμέ χονδρικής, αλλά και στον τελικό καταναλωτή για τη μεταφορά δεδομένων. Γιατί αυτό θα είναι αλλαγή προς όφελος του καταναλωτού και ενδεχομένω στο τέλος ίσως είναι σε θέση ο καταναλωτής κάποια στιγμή να κάνει τις επιλογές του. Σήμερα η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω στους πολίτες που ε, παίρνουν τηλέφωνο είναι όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό να κλείνετε το τηλέφωνό σας. Το καλύτερο πράγμα που μπορώ να τους πω είναι αυτό. Δεν θα πρέπει στη συνένωση όμως να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και διαρθωτικά μέτρα χρειαζόμαστε και ανώτατες τιμές για ε, να υποφελεί ο τελικό καταναλωτή, ο τελικό χρήστη. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα σίγουρα αυτή η προσπάθεια και θα συμμετέχω και εγώ στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Um, thank you very much, uh, Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Κριστιαν Έγκστομ, ευχαριστώ. Συμφωνώ με την συνολικότερη προσέγγιση της Κομισιόν καθώς και με τα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου εδώ. Έχει, ε, δεν, δεν έχει επιτύχει αυτή η προσπάθεια στην αγορά. Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η ρύθμιση. Δεν πρόκειται για την υπόθεση των τηλεπικοινωνιών, για την, για την επιχείρηση των τηλεπικοινωνιών, που είναι σημαντική. Εάν οι επιχειρηματίε δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε αυτέ όταν πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα, είναι αστείο να μιλούμε για ενιαία αγορά. Να πάει ένα επιχειρηματία ε, από τη μια χώρα στην άλλη για να κάνει business και να μην μπορεί να επικοινωνήσει, αυτά δεν είναι σοβαρά. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι, δυστυχώ. Για τις τιμές του τελικού καταναλωτή τώρα για φωνητική, για φωνητική ε, τηλεφωνία και SMS κλπ. Αυτά δεν τα βρίσκω υπερβολικά. Τις τιμές δεν τις βρίσκω υπερβολικές. Όμως, όμως, για την περιαγωγή δεδομένων, δηλαδή για τη μεταφορά δεδομένων σε περιαγωγή, πραγματικά εκεί είναι ε, η, η κατάσταση ε, απίστευτοι πραγματικά καταναλωτές που λαμβάνουν ε, λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ επειδή ξέχασαν να ε, κλείσουν το τηλέφωνο ή να ε, το αποσυνδέσουν από το διαδίκτυο. Αυτές οι ανώτατες οροφές δεν εξυπηρετούν. Αυτές οι τιμές αναφέρονται σε megabyte. Megabyte είναι πάρα πολύ μικρή ε, ποσότητα. Νομίζω ότι δεν χρησιμοποιεί και κανένα ούτω ή άλλω τώρα πια. 1000 MB, δηλαδή ένα GB, αρχίζει και είναι πολύ πιο σημαντικό ως μέτρο. Ο επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης της Ericsson είπε πέρσι ότι ε, θα χρησιμοποιεί ένας καταναλωτής μισό γιγαμπάιτ τον μήνα. Το κόστος παραγωγής ενός μια μεταφορά ενό γιγαβάιτ είναι ένα δολάριο. Ένα ευρώ, πέστε, ένα ευρώ ανά γιγαβάιτ. Οι τιμέ λοιπόν, ενώ η τιμή του καταναλωτή είναι 50 λεπτά ανά μεγαμπάιτ, που μιλάμε δηλαδή για 500 ευρώ το γιγαμπάιτ. Καλά λοιπόν, καλά λοιπόν να βάλουμε αυτά τα price caps, αλλά είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν. Εγώ θα προτείνω λοιπόν από εδώ και μπρο να χρησιμοποιείτε ως μέτρο το gigabyte, που αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, πολύ πιο ενδιαφέρον. Και να εξετάσετε, να, τα πάρετε κάπου σε τάξεις μεγεθών ρεαλιστικές. Έχουμε αυτά τα υπέροχα ευφυή τηλέφωνα τώρα, πραγματικά είναι υπέροχα. Πάρα πολύ χρήσιμα στους καταναλωτές και ακόμα περισσότερο στους επιχειρηματίες. Αν δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Το London Transport έχει μια ε, θαυμάσια εφαρμογή για τα ευφυή τηλέφωνα που είναι όλα τα δρομολόγια μέσα με τις ώρες κτλ. Άχρηστο, άχρηστο. Εάν έχετε ξένη κάρτα SIM, διότι θα σας βγει, βγει πολύ πιο φτηνό να πάρετε το ταξί για να πάτε. Πάνω να κοιτάξετε τα δρομολόγια του London Transport στο ε, ευφύε σας τηλέφωνο. Συμφωνώ και με τους ευρωβουλευτές που μίλησαν πριν και με την Κομισιόν ότι χρειάζονται και δομικές αλλαγές, δομικά στοιχεία και price caps. Αλλά price caps εκεί όπου ανοίγει κάπου η αγορά και προσφέρει δυνατότητες στις επιχειρήσεις και δημιουργούν μια πραγματικά λειτουργική ενιαία αγορά. ας πούμε 10 ευρώ ανά gigabyte. Ένα λεπτό δηλαδή ανά megabyte. Παρ' όλα αυτά θα έχουν οι, οι, πάροχοι των υπηρεσιών αυτών μια, ε, ένα περιθώριο κέρδους της τάξης του 1000%. Ε, πόσο θέλουν τέλο πάντων. Συμφωνώ λοιπόν με τη γενική προσέγγιση, αλλά θα ήθελα να δω να χαμηλώνουν αυτές οι τιμές πραγματικά πολύ πολύ περισσότερο. Σας ευχαριστώ πραγματικά ε, η άποψη ο εμπειρογνώμου. Η κυρία Τούν. Ε, ε, συμφωνώ πολύ με τις προλαλήσαντες. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη χρέωση της περιαγωγής, πώς θα, θα συζητηθεί αυτό και στο μέλλον σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες επιτροπές. Έχουμε ένα πολιτικό-φιλοσοφικό επίπεδο και ένα άλλο τεχνικό το πολιτικό φιλοσοφικό έχει να κάνει με την ενιαία αγορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτή καθ' αυτή, με μια ήπειρο χωρί σύνορα και για την περιαγωγή. Έχουμε αυτή την εικονική πραγματικότητα, αλλά τα ε, σύνορα υπάρχουν στην περιαγωγή και είναι πάρα πολύ οδυνηρά. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική συζήτηση. Την έχουμε την Ενωμένη Ευρώπη επιτέλους ή όχι. Γιατί οι εταιρείε κινητής τηλεφωνίας ε, υψώνουν σύνορα. Και δεν στρέφεται μόνο αυτό κατά της ιδέας της μίας Ευρώπης, αλλά και της ενιαίας αγοράς και της όλης ιδέας του διαδικτύου. Γιατί δεν μπορούμε να ε, αξιοποιούμε, να υποφελούμαστε από όλες τις υπηρεσίες του διαδικτύου που συνέχεια ακούμε να διαφημίζονται. Ε, σύγκριση τιμών, όταν πηγαίνεις σε ένα κατάστημα να μπορείς να χρησιμοποιείς την υπηρεσία αυτή για να συγκρίνεις τιμές. Μήπως είναι πιο φτηνό στη χώρα σου, καλύτερο, δεν ξέρω, το προϊόν αλλά είναι πιο ακριβό να χρησιμοποιήσει κανείς την υπηρεσία από το όφελος που θα είχαμε εάν αλλάξουμε χώρα για να αγοράσουμε ένα προϊόν. Για θέματα ασφαλείας ανατολισμού σε μια πόλη δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εφή τηλέφωνα γιατί μας βγαίνει πανάκριβο. Μόνο το 112 που είναι δωρεάν, αλλά δεν πιάνει και παντού, γιατί το έχω τσεκάρει το καλοκαίρι. Επίσης είμαστε έρμεα των παρόχων. Ανοίγουμε ε, το διαδίκτυο στο ευφυές μας ε, τηλέφωνο και δεν ξέρουμε ποτέ πόσο θα πληρώσουμε, πόσο θα μας χρεώσουν. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο βαριά που πούμε, η πληροφορία, ποια θα είναι η ποιότητα της εικόνας, ε, τι πληροφορίες θα λάβουμε. Έχει ταινία μέσα αυτή η πληροφορία. Αν έχει ταινία είναι καταστροφή. δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει πόσα χρήματα θέλει να δαπανίσει σε αυτή την υπηρεσία. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι προτάσεις που κάνετε, αλλά νομίζω ότι παραμένουν πάρα πολύ περίπλοκες. Μπορεί να έχω γεράσει, αλλά ε, εάν θέλω να ε, επωφεληθώ από την αποσυνδεδεμένη υπηρεσία, να επιλέξω εταιρεία, έχω και άλλες δουλειές. Δεν μπορώ συνέχεια να συγκρίνω τιμές, ποια εταιρεία είναι πιο φτηνή, ποιος πάροχος, ποιο θα διαλέξω κτλ όλα αυτά ε, θα πρέπει να είναι φιλικά προς το χρήστη και τον ε, ε, έτσι, πιο ηλικιωμένο χρήστη εφιών τηλεφώνων. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση και συμφωνούμε όλοι και μας το ζητούν οι πολίτες κινούμαστε όλο και περισσότερο, αγοράζουμε όλα αυτά τα εφή τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και δεν ξέρω τι άλλο. Και όπως γνωρίζετε είναι και η Προεδρία αυτό το καιρό και διοργανώνουμε Ε, μία διάσκεψη με τίτλο «Περιαγωγή χωρίς τέλη περιαγωγής» στις 20 Σεπτεμβρίου. Γιατί παραμένουν τόσο υψηλά τα ε, τέλη περιαγωγής. Το πρωί θα είναι στις 20 Σεπτεμβρίου, 8 και 4 το πρωί παρακαλώ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά και ενδιαφέρουσες και πολύ τολμηρές οι προτάσεις της Πολωνικής Προεδρίας. Σας το έχω στείλει και με email ήδη αυτό και την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές. Ε, απλώς ε, να σας πω ότι θα γίνει και άλλη συζήτηση. Σήμερα συζητάμε τη μελέτη αντικτύπου. Ε, θα συνεχιστεί η συζήτηση ε, για την έκθεση της κυρίας Κόρχολο. Ο καθηγητής Κορέντα Κάμπος. Uh, ε, this, this was αυτή ήταν πολύ καλή παρουσίαση. Εκτιμώ, ε, την εκτίμησα ιδιαίτερα, γιατί έμαθα για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζω και, τώρα, και τόσο καλά. Δεν μιλάμε για μονοπόλιο, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό και όλες οι λύσεις είναι ότι το καλύτερο είναι η προσέγγιση του τομή χειρών βέλτιστων από πολιτικής πλευράς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα. Σας υπενθυμίζω ότι πολλοί οργανώσαμε εκστρατείες στη χώρα μας με βάση τις επιτυχίες που είχαμε στον τομέα της ανώτατης τιμολόγησης της περιαγωγής. Αυτό το χρησιμοποίησαμε σαν βασικό επιχείρημα, γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και η διαφορετικές λύσεις, η διαφορετική λύση φαίνεται αρκετά δελεαστική, αν και είναι δύσκολη. Τουλάχιστον αυτό μας αναφέρθηκε. Ίσως να υπάρχουν και ενδιάμεσες λύσεις που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. in Στις υπηρεσίες υδάτων Υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης προς τον ε, καταναλωτή εάν υπάρχει υπερβολική κατανάλωση νερού, γιατί υπάρχει διαρροή ιδιαίτερα διέτερα κατά, στις περιφέρειες ή ε, σε απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η υποχρέωση και στους παρόχους, δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, εάν η τιμολόγηση είναι πολύ ψηλή Αυτό δεν θα ήταν και ιδιαίτερα δαπανηρό για τους παρόχους. Και υπάρχει και... Έχω και μια τεχνική υφής ερώτηση. Λυπούμε που δεν γνωρίζω το θέμα, αλλά επειδή μιλήσατε για χωριστές χρεώσεις, εγώ έχω ε, δύο αριθμούς και θα εκτιμούσα να έχω έναν. Δηλαδή να έχω το, την ίδια SIM και την ίδια σύσκευη, το ίδιο τηλέφωνο. Με βάση την, τις χωριστές χρεώσεις από τεχνικής πλευράς θα ήταν εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Ή υπάρχει λόγος γιατί είναι δύσκολο κάτι τέτοιο να γίνει χωριστή χρέωση με την ίδια ΣΥΜ. Κύριε Ρόιτοβα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση και να επανέλθω λίγο στο ιστορικό της υπόθεσης. Πριν από μία πενταετία συζητούσαμε πάρα πολύ σοβαρά εάν μπορούμε καν να ρυθμίσουμε ε, τις ε, τιμές και τις υπηρεσίες περιαγωγής και τη δημολόγησή τους. Και τότε μας έλεγαν οι εταιρείε της ε, τηλεφωνίας ότι αν ε, εισαγάγαμε ανώτατες τιμές θα έπαιρναν πίσω τα χρήματα που θα έχαναν από άλλες υπηρεσίες. Εσείς το έχετε αναλύσει αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε δει να αυξάνουν τις τιμές αλλού οι πάροχοι ε, στην υπηρεσία δεδομένων από το διαδίκτυο ή όχι. Και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι αν βάλουμε ανώτατε τιμέ θα πτώχευαν, πώ αντέδρασαν και ποια είναι η κατάστασή του Και ένα δεύτερο, μια εμπειρία μου. Τώρα η αγορά είναι υποχρεωμένη ε, σε κάποια δράση ε, στη μεταφορά δεδομένων ADSL. Στη Τσεχική Δημοκρατία χρειαζόμαστε πέντε εβδομάδες για να αλλάξουμε πάροχο. Εγώ το, ε, το αυτό όταν θέλησα να αλλάξω εταιρεία και δεν είμαι η μοναδική. Ένα τρίτο. Εχθές άνοιξα το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο εδώ στις Βρυξέλλες Μάλλον άνοιξα το γραμματοκιβώτιό και ανακάλυψα ότι έχει αυξηθεί η τιμή στην τηλεφωνία, την κινητή και στο διαδίκτυο ε, χωρίς να με ρωτήσουν. Μου λένε υποτίθεται ότι θα είναι καλύτερη η ε, παροχή υπηρεσίας, ότι θα έχω καλύτερο διαδίκτυο, αλλά έβαλα να δω τσεχική τηλεόραση και δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Μάλλον έχει επιδεινωθεί η ποιότητα. Ε, Χρειάζεται μια ανάλυση λοιπόν των όσων συμβαίνουν στην πραγματικότητα και τι κάνουν οι πάροχοι ε, όταν υποτίθεται ότι αναβαθμίζουν το δίκτυο ή απελευθερώνονται από άλλους παρόχους και τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές από ε, μπελάδες και προβλήματα. Τελικά εγώ έχω την εμπειρία ότι κάποιο επιστρέφει στην αρχική του εταιρεία γιατί δεν έχει ούτε το κουράγιο, ούτε το χρόνο, ούτε τα ε, χρήματα, ούτε τη διάθεση τελικά να ψάχνει παραπονέθηκα, αλλά ε, διαπίστωσα ότι ορισμένοι ούτε καν αυτό δεν κάνουν. Και τώρα τι γίνεται με το ψηφιακό περιβάλλον για τους επιχειρηματίες. Ε, η περιεγωγή είναι πολύ πιο σημαντική ε, στα δεδομένα από ότι τα SMS. Τώρα λέμε ότι θα λύσουμε διάφορα θέματα το 2015. Αυτό είναι πολύ αργά όμως. Μας προσπερνούν οι εξελίξεις στην αγορά ε, κανονικά εμείς θα πρέπει να προηγούμαστε και να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις και να τις προκαλούμε. Γιατί τα λέω όλα αυτά, τι θέλω να πω. Ο όγκος των χρημάτων για τη μεταφορά δεδομένων οφείλεται το γεγονός ότι δεν ξέρουν πόσο θα τους κοστίσει ε, στο τέλος του μήνα. Δεν, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές οι καταναλωτές μεταφοράς δεδομένων από το τηλέφωνο γιατί δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν. Αν ξέρουν, αν είναι ενήμεροι, μπορεί να χρησιμοποιούν περισσότερο αυτές τις υπηρεσίες και τελικά να μειωθεί η τιμή. Καλωσορίζω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι το σημαντικότερο στοιχείο εδώ δεν είναι η οροφή στη τιμολόγηση, αλλά να εξηγήσουμε εκ των προτέρων στους καταναλωτές πριν χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία πόσο αυτή κοστίζει. Αυτό το ίδιο που γίνεται και με τη φωνητική τηλεφωνία και την περιαγωγή. Να μπορεί ε, ο καθένα να συγκρίνει τιμές σε μια ιστοσελίδα μεταξύ διαφόρων παρόχων και να ξέρουμε ότι η μια εταιρεία χρεώνει το gigabyte τόσο, η άλλη τόσο. Να το γνωρίζω εκ των προτέρων όμω πόσο θα μου κοστίσει. Αν θα ανοίξω το smartphone αυτό ε, θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε ως υπηρεσία. Να πω κι εγώ λίγα πράγματα, κυρίως ε, στην κατεύθυνση της κυρίας Ρόιτοβα. Αυτά που λέτε υπάρχουν. Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν σας προσφέρει αυτές τις προφορίες, τότε δεν σέβεται τις υποχρεώσεις που έχουμε θεσπίσει εμείς ως ε, κοινοβούλιο. Εδώ στο δικό μου λέει καθαρά πόσο θα σας κοστίσει να έχετε διαδίκτυο, να έχετε περιαγωγή, να στείλετε ένα SMS. Τα έχουμε αυτά τα πράγματα ήδη. Και απαντώντας τον κύριο Ντεκάμπος, πάλι μετά από δική μας πρόταση και λόγω του σοκ που έχουν πάθει πολλοί καταναλωτές ε, έχουμε βάλει ένα ανώτατο όριο που υποτίθεται ότι θεσπίζουν, βάζουν οι, οι υπηρεσιών στα 15 ΜΜ. Βεβαίως πρόκειται σήμερα για μια αφετηρία και ούτε επικρίνω κανένα. Αλλά ας γνωρίζουμε τι ήδη διαθέτουμε. Και πολλά από αυτά ξεκίνησαν από ιδέες της δικής μας Επιτροπής. Μην υποτιμάτε τα όσα έχουμε επιτύχει δηλαδή. Εάν δεν έχετε αυτές τις πληροφορίες, τότε δεν συμμορφώνεται ο πάροχος υπηρεσιών σας με τις, ε, με τις ε, υποχρώσεις του. Ας διαβάζετε λοιπόν πρώτα τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Γεγονός είναι λοιπόν τώρα ότι με την επόμενη γενιά ευφυών τηλεφώνων γίνεται όλο και πιο εύκολη η πρόσβαση στα δεδομένα. Και Βεβαίως είναι πιο εύχριστα τα τηλέφωνα αυτά και ε, μπορούν πολύ πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ούτω καθεξής και αυτά τα συνηθίζουμε. Το παράδοξο είναι ότι αυτά λειτουργούν στο εγχώριο δίκτυο. Αν όμως πάτε στην Αλοδαπή, στη χώρα μου τουλάχιστον, και κλείστε το τηλέφωνο, οι περισσότεροι θέλουν ένα, ε, μια υπηρεσία που να έχει μια χρέωση κατά αποκοπή και εγώ εξέτασα σε μια πολύ απλή εφαρμογή την ώρα που σας μιλούσα πόσα δεδομένα χρησιμοποίησα στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορώ να έχω την πληροφορία αυτή μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν ανησυχώ λοιπόν. Αυτή τη στιγμή όμως εξέλθω του Ηνωμένου Βασιλείου, κλείνω την περιαγωγή ε, δεδομένων μου. Και αν σκεφτείτε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, πώς έχουμε φτάσει δηλαδή όπου όλοι αυτοί επενδύουν στην εύχρηστη περιαγωγή δεδομένων. παρόλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμό στην αγορά, δεν επωφελείται τελικά ο καταναλωτή. Και αυτό έχει δίκιο ε, η κυρία Ροϊδοβά. Και ένα από τα προβλήματα που έχουμε με τι προτάσει περιορισμού των τιμών, και που είναι πολύ τεχνικέ βέβαια, εμεί είμαστε εκείνοι, πιστεύω, μέσα ναι, στη συζήτηση αυτή που θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν για να τα κάνουμε αυτά πιο εύχριστα για τον καταναλωτή. Για το άμεσο μέλλον μέχρι το 2015 το πρόβλημα είναι ότι οι διαθωτικές αλλαγές προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικές ως προσπάθεια επίλυση του προβλήματος, αλλά δεν έχω την εντύπωση, ίσως βέβαια να μην προλάβει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δέχονται ότι δεν έχουν σκεφτεί και πολύ σε βάθος. Οι Μπέρεκ που είναι οι ε, ε, Ευρωπαίοι ρυθμιστές ε, της κινητής τηλεφωνίας έκαναν προτάσεις και, και ήδη αμφισβητούν τις, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 300 εκατομμυρίων που είπε προηγουμένως δεν ξέρουμε τελικά ποιο θα είναι το κόστος, ούτε ξέρουμε αν θα είναι τεχνικά εφικτό, ούτε ξέρουμε αν θα είναι και εύχριστο. Εγώ θεωρώ ότι η διαρθρωτική λύση είναι μεν σημαντική, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά για τις ε, διαρθρωτικές αυτέ λύσει. και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο σε μια παράταση και ε, και ένα πιο ε, και ένα σφίξιμο των οροφών των τιμών ε, να οδηγηθούμε έτσι σε περισσότερο ανταγωνισμό, γιατί το πρόβλημα, κύριε Δεκάμπος, δεν είναι μονοπόλιο, αλλά ότι ολόκληρη η δομή της αγοράς, γιατί υπάρχουν πολλοί πάροχοι υπηρεσιών, δεν επιτρέπει τον ανταγωνισμό. Όμως, εν τέλει, πόσοι καταναλωτές πραγματικά ψάχνουν να βρουν τις φθηνότερες επιλογές. Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να πιεστούν οι ίδιοι οι πάροχοι υπηρεσιών να προσφέρουν πιο ελκυστικά πακέτα. Αυτό βέβαια ήδη γίνεται. Εδώ ε, διάβασα ότι θα έχω 3 λίρες ανά μεγαμπάιτ για να κατεβάσω δεδομένα. Και εδώ μου λέει ότι άλλο, ε, άλλη επιλογή είναι 30 MB την ημέρα για 3, για 3 λίρες. Αυτά λοιπόν τα πράγματα ήδη γίνονται ε, στην αγορά ήδη και τι πληροφορίες αυτέ τι λαμβάνετε και στο κινητό σα τηλέφωνο. Λοιπόν, το έργο που μας αναμένει είναι ενδιαφέρον. Η προσέγγιση μα είναι βεβαίω υπέρ του συμφέροντος των καταναλωτών. Το impact assessment της Κομισιόν είναι σημαντική αφετηρία και το δικό μου πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι βασικέ διαρθρώσεις που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να διατηρήσει τις ε, ε, οροφέ των τιμών κλπ, είναι καταρχήν σωστά. Εγώ νομίζω ότι οι διαθωτικές αυτές ε, αλλαγές είναι σωστές και θα περιμένουμε και την έκθεση της Μπέρεκ και να προσκαλέσουμε και τον πρόεδρο της Μπέρεκ, των Ευρωπαίων δηλαδή ρυθμιστών, να, έρθουν να έρθει εδώ να μας εξηγήσει τις απόψεις τους. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να προσκαλέσω τον πρόεδρο της Μπέρεκ να έρθει εδώ στην Επιτροπή να μας μιλήσει όχι μόνο για την περιαγωγή αλλά και για άλλα θέματα καταναλωτών. Και πώς τα στοιχεία προστασίας των συμφερόντων καταναλωτών εφαρμόζονται στην πράξη στις χώρες μέλη. Γιατί πολλά από τα όσα είπατε τώρα, δηλαδή η δυνατότητα της κυρίας Ρόιτοβα να αλλάξει παρόχους υπηρεσιών, οι αλλαγές όρων, η προσυμβατική ενημέρωση, τα πράγματα για τα οποία παραπονείστε καλύπτονται, καλύπτονται στο πακέτο το οποίο έφτιαξε η Επιτροπή μας. Ε, μάλιστα εγώ ήμουν εισηγητής. Ας πάρει κυρία Ρόιτοβα τον φάκελό μου που είχα φτιάξει και να πάει στον πάροχο υπηρεσιών και να του πει κοιτάξτε γιατί δεν συμμορφώνεστε με αυτά που έχει ε, αποφασίσει, εγκρίνει και επιβάλλει η Επιτροπή μου. Το πρόβλημα νομίζω είναι ότι δεν συνεργαζόμαστε αρκετά με τους εθνικούς ρυθμιστές για να φροντίσουμε να εφαρμόζονται τα όσα έχουμε αποφασίσει εδώ. Λοιπόν, χρειάζεται να σκεφτούμε λίγο περισσότερο και μάλιστα προς τα πρόσωπα θα έλεγα, προς το μέλλον δηλαδή, το γεγονός ότι βέβαια η μεταφορά δεδομένων σε περιαγωγή θα είναι κυρίως ο τομέας εκείνος αγοράς που θα αναπτυχθεί περισσότερο. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ και τον κύριο Κόρχολα. Θα ήθελα παρακαλώ να σας δώσω δύο λεπτά, αν θέλετε να επανέλθετε. Βέβαια θα επανέλθετε και αργότερα για να μας απαντήσετε. Μετά όμως να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, ορισμένα ε, γενικά ζητήματα που θα ήθελα να θίξω. Ε, τέθη ένα ερώτημα κατά πόσο οι πολίτες θα επιλέξουν εναλλακτικέ προσφορές περιαγωγής, αν είναι διαθέσιμες και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι περίπλοκο, εάν υπάρχει αυτό το φάσμα επιλογών. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα δίλημα. Εάν δεν υπήρχε επιλογή, θα ήταν εύκολο να διαλέξετε τον πάροχο και δεν θα είχατε πολλά πακέτα επιλογής. Όμως, δεν θα υπήρχε ούτε ανταγωνισμός. Αν έχετε περισσότερες επιλογές υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε μια εξισορρόπηση των δύο αυτών στόχων. Δηλαδή να υπάρχουν προσφορές που είναι ανταγωνιστικές και να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή αυτό βεβαίως θα πρέπει να το κάνουμε κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχουν επιλογές για τον καταναλωτή κατά εύκολο τρόπο, με εύκολο τρόπο για εκείνους που θέλουν να συγκρίνουν τιμές και αυτοί που θέλουν να βρουν ενδιαφέρουσες προσφορές, βεβαίως δεν περιμένουμε από κάθε καταναλωτή να ελέγξει τις εναλλακτικέ, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχουν. Εάν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα καταναλωτών που συντρίνει τιμές, που επιλέγει πάροχο σύμφωνα με τις τιμές, τις διαθέσιμες τιμές, τότε εάν υπάρχει επαρκές ποσοστό αυτό οδηγεί σε ανταγωνισμό στην αγορά και προωθεί τους παρόχους, οθεί τους παρόχους να μειώσουν τις τιμές. Δεν σημαίνει ότι κάθε καταναλωτής πρέπει να το κάνει αυτό, απλώς θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους καταναλωτές που προβαίνουν σε τέτοιες συγκρίσεις. Επίσης θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω ως προς την ε, κατανάλωση ε, δεδομένων. Υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση, υπάρχουν όλο ένα και περισσότεροι που συγκρίνουν τις τιμές. Και αν υπήρχε μια εναλλακτική προσφορά, δηλαδή ε, μια προσφορά που θα ήταν διαφανής και θα διαφημίζεται σωστά, τότε θα μπορούσε να ευεργετηθεί ολόκληρη αγορά. Τώρα κατά πόσο η διαρθρωτική λύση είναι εφικτή από τεχνικής πλευράς. Βεβαίως στον τομέα της ε, μηχανικής όλα είναι εφικτά και με βάση ε, τα στοιχεία ανάδρασης από την βιομηχανία βλέπουμε ότι αυτή είναι μία από τις λύσεις. Υπάρχουν άλλες λύσεις που είναι λιγότερο δαπανηρές, που είναι ε, πιο ε, εφάρμοστες. Εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Εάν υπάρχει λοιπόν εναλλακτική, θα πρέπει να διευκολύνει την επιλογή. έτσι ώστε οι πάροχοι να μπορούν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Τέλος, ως προς τη μεταφορά δεδομένων μέσω περιαγωγής και την ανώτατη τιμολόγηση, εάν θέλουμε να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα για να μπορεί κανείς να μπει στην αγορά. Εάν η τιμολόγηση είναι χαμηλή, τότε οι καταναλωτές θα δεχτούν αυτές τις κατά Και αυτό είναι πολύ καλό για τον καταναλωτή, τη στιγμή που υπάρχουν ρυθμισμένες τιμολογήσει. Αλλά όπως είπε και η απόφαση του ΔΕΚ, η ρύθμιση των τιμών θα πρέπει να έχει προσωρινή μορφή, να ισχύει προσωρινά. Δηλαδή δεν μπορούμε να βασιστούμε στη ρύθμιση τιμών στο δίνεκες. Ως προς την τιμολόγηση μεταφοράς δεδομένων, φυσικά πρόκειται για ένα κόστος που είναι ψηλότερο από αυτό της ανώτερης, ανώτατης τιμολόγησης, αλλά θα πρέπει να ε, μας απασχολήσει σε σχέση με τα SMS. Πρόκειται για μια αγορά η οποία ένα και εξελίσσεται. Δεν θα πρέπει να στρεβλώσουμε την αγορά. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες προσφορές ήδη διαθέσιμες και θα πρέπει να παροτρύνουμε τους παρόχους να μας προβάλλουν δελεαστικότερες προσφορές. Η διαδικασία αυτή ανταγωνισμού θα μειώσει τις τιμές ε, στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εισήγηση και αυτή η συζήτηση, η προκαταρκτική συζήτηση. Η κυρία Κορχόλα θα ε, το προθίσει το ζήτημα αυτό στην έκθεσή της και θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων πριν γίνει αυτό. Θα συζητήσουμε και το χρονοδιάγραμμα εγκαίρως και στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Θέλετε κάτι να πείτε εν κατακλείδη, ναι, λίγα λόγια επειδή είμαι Φινλανδή ε, δεν μιλώ ε, μακρόν συνήθως. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ ε, για τις απογοητεύσεις που μας αναφέρατε και που ζείτε στο εξωτερικό. Τι υπηρεσίες έχουμε πραγματικά ο κύριος Δεκάμπος έδειξε ένα πολύ σωστό θέμα, διότι έχω μία υπηρεσία που με πληροφορεί ε, όταν ε, βρίσκομαι στο εξωτερικό, αλλά δεν ξέρω ποιο ε, είναι, πώς λειτουργεί η μεταφορά δεδομένων και ποιο είναι το συνολικό κόστος. Εγώ έχω το σύστημα προειδοποίησης στο τηλέφωνο μου, αλλά δεν είναι επιγραμμικό το σύστημα όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό, δηλαδή τα στοιχεία τα βλέπω μετά. Αυτό πραγματικά ισχύει, δηλαδή εκτός ε, παρόχου, δηλαδή εκτός εθνικού παρόχου δεν λειτουργεί το σύστημα online στην Αλλοδαπή γιατί εκεί που χρειαζόμαστε χάρτες και χρονοδιαγράμματα, τα χρειαζόμαστε στην αλλοδαπή. Μπορούμε να τα με το FES τηλέφωνο, αλλά είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το δείτε με το προμηθευτή σας. Το πάροχο. Ε, γιατί δεν απολαμβάνετε των δικαιωμάτων που δικαιούστε και που σας έχουμε εμείς ε, ε, εξασφαλίσει. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη ε, από τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας και Προστασίας των Καταναλωτών να μας παρουσιάσουν τα πολύ ενδιαφέροντα που μελετούν για την συνειδητοποίηση των καταναλωτών. You have copies Ενίσχυση του ρόλους. Ε, μπορείτε να μας παρουσιάσετε σε συντομία, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, τα συμπεράσματά σας. Έχετε τον υπολογιστή, παρακαλώ. Να το χειριστείτε μόνοι σας. Σας δώσω το λόγο. Είμαστε έτοιμοι τώρα και οι διαφάνειες ε, στις οθόνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θα συντομεύσω την παρουσίασή μου, θα σας δείξω λιγότερες διαφάνειες από εκείνες που έχετε στην τυπωμένη ε, έκδοση. To present ε, θέλω να ε, σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη για την ενίσχυση του ρόλου του καταναλωτού. Γιατί κάναμε αυτή τη μελέτη, την έρευνα. Έχουμε μια στρατηγική ενίσχυση του ρόλου και συνειδητοποίηση των καταναλωτών. Γιατί ένα ενήμερο καταναλωτή με δύναμη παίρνει τι αποφάσει που τον αφορούν. Ε, κοιτάει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ε, τα αντιμετωπίζει με καλύτερο τρόπο και ενισχύει και τον ανταγωνισμό και την καινοτομία και τελικά είναι πιο ανταγωνιστικές, πιο καινοτόμες και πιο ειλικρινείς οι εταιρείε. Πριν κάνουμε αυτή τη μελέτη δεν υπήρχαν συλλογικά στοιχεία ολοκληρωμένα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και το ρόλο τους. Με την παρούσα μελέτη καταλαβαίνουμε καλύτερα τους καταναλωτές και γνωρίζουμε περισσότερο ε, τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές και τι είναι πρόθυμοι να κάνουν. Έτσι ε, θα ρυθμίζουμε καλύτερα, θα κανονίζουμε καλύτερα την αγορά και θα ε, παίρνουμε καλύτερες πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είναι σημαντικό και για μας αλλά και για τα κράτη-μέλη που παίρνουν εθνικές αποφάσεις. Λοιπόν, έγινε αυτή η μελέτη πότε πέρυσι, συνεργαστήκαμε με τη Eurostat 55.000 ε, καταναλωτές συμμετείχαν σε 27 κράτη-μέλη, ε, στην η Νορβηγία και την Ισλανδία. 55.000 είναι πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Κοιτάξαμε και μεταβλητές κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα όπως είναι η ηλικία, η μόρφωση, η χρήση του διαδικτύου για να εκτιμήσουμε ποιες είναι εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που μπορεί να είναι πιο ευάλωτες ως καταναλωτές από κάποιες άλλες. Τα βασικά ζητήματα που μας απασχόλησαν στη μελέτη αυτή ήταν η εμπιστοσύνη ε, που έχουν για τους αυτούς τους καταναλωτές ε, στις δυνατότητές τους, οι δυνατότητες να διαβάζουν ε, λογοτύπους, ετικέτες, να λογαριάζουν τις τιμές, να γνωρίζουν την νομοθεσία υπέρ τους και συμπεριφορά των καταναλωτών, συμμετοχή των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά σύγκριση τιμών, να διαβάζουν όρους ε, ε, και ετικέτες και αν ενδιαφέρονται για την ενημέρωσή τους ε, και τι εμπειρία έχουν στην αγορά προϊόντων. Επίσης, τι δράσεις είναι πρόθυμοι να αναλάβουν όταν έχουν προβλήματα με καταγγελίες, με παράπονα ε, σε ένα κατάστημα ή άλλο. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω σε αυτά τα πέντε βασικά κεφάλαια τα ευρήματά μας και τις ερωτήσεις που κάναμε για να καταλάβετε ακριβώς ε, τι ε, ρωτήσαμε τους καταναλωτές και τι ζητήσαμε με αυτούς. πρώτο η εμπιστοσύνη που έχουν στον εαυτό τους αυτοπεποίθηση όταν αγοράζουν κάτι. Δηλαδή, ε, είναι συνειδητοποιημένοι οι καταναλωτές, καταλαβαίνουν τι κάνουν εκείνη την ώρα και πόσο καλά θεωρούν ότι προστατεύονται από το δίκαιο για τους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντική η αντίληψη που έχει ο καθένας για τον εαυτό του ως καταναλωτή. Γιατί ένας συνειδητοποιημένος καταναλωτής έχει και περισσότερες ικανότητες και περισσότερες δυνατότητες. Ε, ευρήματα. 73% των καταναλωτών έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 63% θεωρούν ότι γνωρίζουν και 55% ότι προστατεύονται. Αλλά μόλις 44% των απαντήσεων έλεγαν και τα τρία στοιχεία ταυτόχρονα, ότι ήταν και συνειδητοποιημένοι και ε, ενήμεροι και προστατευμένοι, ενώ 17% κανένα από τα τρία. Επίσης, Κάτι άλλο που θα δούμε σε όλη τη διάρκεια της μελέτης είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή σε πέντε χώρες 20% ή λιγότερο των απαντήσεων είχαν και τα τρία στοιχεία αυτά της εμπιστοσύνης, της γνώσης και της προστασίας. Αν δούμε το κοινωνικό-οικονομικό σκέλος, διαπιστώνουμε ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη και με την ηλικία αυξάνεται με τη μόρφωση και οι χρήστε του διαδικτύου έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στι δυνάμεις του. Ε, το επόμενο που μελετήσαμε είναι οι ικανότητε ε, των ε, καταναλωτών αν μπορούν να διαβάζουν λογοτύπους, ετικέτε και να κάνουν μαθηματικές πράξεις, αριθμητικές. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάναμε. Για να καταλάβουμε αν οι καταναλωτές είναι σε θέση να καταλάβουν και να πάρουν μια απόφαση αγοράς. Ερώτηση πρώτη. Η ίδια ε, τηλεόραση ε, πωλείται στο κατάστημα Α και στο κατάστημα Β. Ποια είναι πιο φτηνή. Στο κατάστημα Α κάνει 500 ευρώ με 10% έπτωση. Και στο δεύτερο κατάστημα ε, κοστίζει 400 ευρώ. Προφανώς η πιο φθηνή τηλεόραση είναι στο β' κατάστημα. Μόνο το 20% των ε, καταναλωτών ε, έδωσαν λάθος απάντηση σε κάτι που οι περισσότεροι από εσάς θα θεωρείτε πάρα πολύ απλό υπολογισμό. Σε ορισμένε χώρες ε, έφταναν και το 30% και το 40% εκείνοι που δεν μπορούσαν να απαντήσουν σωστά σε αυτή την ερώτηση. Similar, uh, sort of percent... λοιπόν, ε, ό,τι αφορά τα ποσοστά, επόμενη ερώτηση σε ό,τι αφορά ένα λογαριασμό, αποταμίευση, τράπεζα, ε, καταθέσεων, ε, ποιο ήταν ε, το καλύτερο επιτόκιο, το πιο ενδιαφέρον, 1, 2, 3, 4%. Και πάλι το 20% των απαντήσεων των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη ήταν λάθος. Και σε μερικά κράτη-μέλη έφταναν και μέχρι το 40%. The last question that I want... Επόμενη ερώτηση. Και πάλι ε, το τόκο. Αν ε, κάποιος έχει ένα δάνειο 50.000 ε, με τόκο 6, ε, επιτόκιο 6% πόσο τόκο θα πληρώσει για τον πρώτο χρόνο. Βεβαίως είναι 3.000 ευρώ η απάντηση. 56% ήταν οι σωστές απαντήσεις για το πρώτο έτος ότι είναι 3.000 ευρώ ε, ο τόκος. Το 25% των απαντήσεων ήταν δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και οι υπόλοιποι απάντησαν λάθος. Σε ορισμένες χώρες, πάνω από τους μισούς καταναλωτές είπαν ότι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Συμπέρασμα των τριών αυτών ερωτήσεων. Λιγότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά και στις τρεις ερωτήσεις. 34% έχουν ε, δύο σωστές απαντήσεις, 15% ε, μία και 6% καμία από τις τρεις ερωτήσεις δεν απάντησαν σωστά και να δούμε ε, κοινωνικά και τα δημογραφικά. Ηλικία 25 ε, ε, με 54 είναι η ηλικία που δίνει τις πιο σωστές απαντήσεις. Δηλαδή οι πιο νεαροί και πιο ηλικιωμένοι καταναλωτές απαντούσαν λάθος. Επίσης, ελέγξαμε κατά πόσο γνωρίζουν λογοτύπους. Ρωτήσαμε ε, τους δείξαμε διάφορους λογοτύπους και τους ρωτήσαμε, τους γνωρίζετε, τους έχετε ξαναδεί και τι σημαίνουν αυτοί. Πέντε τους δείξαμε συνολικά, ένας είναι ε, αυτός αυτό σημαίνει βεβαίως ότι το προϊόν ε, ανταποκρίνεται στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έξι ήταν κάθε φορά οι απαντήσεις για κάθε ένα από τους λογοτύπους. Αυτό το γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι. 66% είπαν ότι γνώριζαν αυτό το λογότυπο. Όταν τους ρωτήσαμε όμως τι σημαίνει, ποια ήταν η σωστή ερμηνεία, οι περισσότεροι απάντησαν λάθος. Ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόλις 25% απάντησαν σωστά ότι η απάντηση είναι ε, ότι είναι σύνομο με την κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εδώ βλέπετε και τους υπόλοιπους λογοτύπους που δείξαμε. Το πρώτο είναι προϊόν βιολογικής γεωργίας, μετά ε, αυτό που σας είπα προηγουμένως για το ΣΥΗ. E, το τρίτο είναι, ανταποκρίνεται σε αυστηρές οικολογικές προδιαγραφές το τέταρτο από χαρτί που ανακυκλώνεται προϊόν και το τελευταίο ένα προϊόν που μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία σας. Και βλέπετε κάθε φορά πόσο γνωρίζει ο κόσμος αυτά τα σήματα, τους, τα σύμβολα, την βιολογική γεωργία και τις οικολογικές προδιαγραφές δεν τη γνωρίζουν, ενώ στη δεύτερη στήλη βλέπετε πόσοι απάντησαν σωστά ως προς τη σημασία αυτού του λογοτύπου γενικά διαπιστώσαμε ότι πάνω από το 1 πέμπτον των όσων απάντησαν δεν μπορούσαν να ε, απαντήσουν σωστά για κανένα λογότυπο. Και μόλις 2% τα γνώριζε όλα. επόμενος τομέας που μελετήσαμε ήταν η γνώση των καταναλωτών της νομοθεσίας. Ε, κοιτάξαμε και ε, ελέγξαμε εάν γνωρίζουν τα τι, τι ισχύει για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, για τις ε, περιόδους περισυλλογής και αλλαγής γνώμης και για τις εγγύησεις. Του ρωτήσαμε. Σα στέλνουμε το ταχυδρομείο δύο DVD εκπαιδευτική τηλεόραση που δεν ε, παραγγείλατε μαζί με ένα λογαριασμό 50 ευρώ. Είστε υποχρεωμένο να πληρώσετε το λογαριασμό. Η απάντηση είναι όχι. Και επίση δεν είστε υποχρεωμένοι να στείλετε πίσω τα DVD. Λιγότεροι από 4 στου 10 απάντησαν σωστά. Συγκεκριμένα 39%. Πάνω από τους μισούς θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν το λογαριασμό μένα, αλλά πρέπει να στείλουν πίσω τα DVD. Επόμενη ερώτηση. Ε, για τις διαφημίσεις για τις τιμές. Ποιος ε, κανόνας νομίζετε ότι ισχύει για τη διαφήμιση τιμών αεροπορικών εισιτήριων. Η απάντηση βεβαίως η σωστή είναι η πρώτη. Θα πρέπει η διαφήμιση να περιλαμβάνει τη τιμή συνολικά, μαζί με τέλη, ε, φόρους κτλ. Μόνο 56% απάντησα σωστά ότι θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό ποσό και τα τέλη αεροδρομίου και ε, διάφορες επιβαρύνσεις και φόροι. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση γιατί ήταν η μοναδική όπου οι καταναλωτές στις βόρειοευρωπαϊκές χώρες που συνήθως απαντούν σωστά απάντησαν λάθος. Γιατί πολλοί συστά μας είπαν ότι ε, ε, η σωστή απάντηση είναι η 2 ή η 3. Ή ότι δεν υπάρχει ειδικό κανόνα ή ε, δεν ήταν υποχρεωμένη η αεροπορική εταιρεία να συμπεριλάβει και τα τέλη παρά μόνο το κόστος της πτήσης. Και τέλος, μια ερώτηση για την εγγύηση του προϊόντος. Φανταστείτε ότι αγοράσετε ένα νέο ψυγείο καινούριο πριν από 1,5 χρόνο, χάλασε, δεν πήρατε επιπλέον εμπορική εγγύηση, ε, είναι μέσα στην εγγύηση ε, η δωρεάν επισκευή. Βεβαίως, ναι είναι η απάντηση γιατί είναι διετία. Μόνο 39% απάντησαν σωστά και ξέρουν ότι ε, μέσα σε μια διετία ε, δικαιούνται δωρεάν επισκευή αντικατάσταση του ψυγείου. Από την άλλη, 44% θεωρούν ότι έχει λήξει η εγγύηση. If, if, you look at uh, consumer awareness... Εάν δούμε λοιπόν τη συνειδητοποίηση και των 7 ερωτήσεων που κάναμε στους καταναλωτές για τη νομοθεσία υπέρ καταναλωτών, μόλις 2% απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Και ε, αντίστροφα 4% απάντησα λάθος σε όλες τις ερωτήσεις. Η Γερμανία και η Φιλανδία είχαν τις καλύτερες επιδόσεις, αλλά η Νορβηγία ήταν ακόμα καλύτερη, ακόμα και από τη Γερμανία και τη Φιλανδία. Από όλες τις χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης ε, οι καταναλωτές που είναι και πιο ενήμεροι και πιο συνειδητοποιημένοι και ε, γνωρίζουν για την προστασία τους, δίνουν τις καλύτερες απαντήσεις. Θα σας δώσω μόλις ε, λίγα στοιχεία, ευρήματα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών ε, οι γυναίκες βεβαίως ε, πηγαίνουν περισσότερο στην αγορά από τους άνδρες, δύο ώρες την εβδομάδα. 49% γνωρίζουν για μια οργάνωση προστασίας καταναλωτών. Πάνω από 6 στους 10 έχουν δει μια φορά στη ζωή τους ένα πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών. Μόλις 17% κάθε εβδομάδα Όποιος γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά του, διαβάζει ε, για την προστασία των καταναλωτών ή βλέπει στη τηλεόραση αντίστοιχα προγράμματα. Και τέλος, μιλούν οι καταναλωτές σε άλλους καταναλωτές για την εμπειρία τους και ε, μοιράζονται μάλλον τις θετικές εμπειρίες τους παρά τις αρνητικές. Το τελευταίο στομέα που μελετήσαμε ε, είναι τα προβλήματα που έχουν οι καταναλωτές και η προθυμία τους να αναλάβουν κάποια δράση και η δυσαρέσκειά τους. Μετρήσαμε λοιπόν ότι ένας στους πέντε καταναλωτές μας δήλωσε πρόβλημα με ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ένα πάροχο λιανικής ε, το περασμένο έτος και θεωρούν ότι δικαιούνται να διαμαρτυρηθούν. Αν δείτε τη διαφάνεια, από όσου δήλωσαν πρόβλημα το 63% είπαν ότι είχαν ένα πρόβλημα και μόνο, ενώ ε, λιγότεροι είπαν ότι είχαν περισσότερα προβλήματα. Κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι όσο καλύτερα γνωρίζουν ε, τα δικαιώματά τους οι καταναλωτές τόσο περισσότερο δηλώνουν και το πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα προβλήματα αλλά δεν τα αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές γιατί δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους. Επίσης, ζητήσαμε από τους καταναλωτές να υπολογίσουν την οικονομική του ζημία και κατά μέσο όρο είναι 374 ευρώ. Αυτό όμως επηρεάζεται από λίγους καταναλωτές που έχουν δηλώσει πάρα πολύ μεγάλες ζημίες. Οι περισσότεροι ε, δηλώνουν 20 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Από εκείνους τους καταναλωτές λοιπόν που είχαν πρόβλημα, τα τρία τέταρτα ανέλαβαν κάποια δράση, προσπάθησαν να αποζημιωθούν για την απώλεια. Και οι περισσότεροι απευθύνθηκαν στο κατάστημα ή στον πάροχο λιανικής. Και πολύ λίγοι ήταν οι καταναλωτές που προχώρησαν σε πιο επίσημη δράση. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη που δείχνει πόσο συνειδητοποιημένοι είναι οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες για το ρόλο τους και τη δύναμη που έχουν. Ε, έχουμε και ένα δείκτη ε, που έχει να κάνει με τις δυνατότητες, τη γνώση των δικαιωμάτων τους και τη ε, δράση συμμετοχή των καταναλωτών. Οι πιο ισχυρέ χώρε εδώ είναι η Νορβηγία που γενικά έχει τι καλύτερε επιδόσει παντού. Φιλανδία, κάτω χώρε, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Αυστρία και Ισλανδία. Αυτές είναι οι χώρες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Στη μέση είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, ε, το Ενό Βασίλειο, η Κύπρο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Μάλτα. Και ε, οι υπόλοιπε χώρες είναι πιο κάτω στην κλίμακα. Αν σας ενδιαφέρει η χώρα σας, κοιτάξτε τη λεπτομερή έκθεση γιατί θα δείτε πολύ περισσότερα στοιχεία εκεί. Ε, θα διαπιστώσετε ότι οι καταναλωτές διαφέρουν στις συμπεριφορές από χώρα σε χώρα, αλλού γνωρίζουν περισσότερα, αλλού μπορούν περισσότερα. Και αυτός ο, ο ε, ε, είναι σε ευθεία σχέση με το εισόδημα και το ΑΕΠ της χώρας. Λοιπόν, τι συνέχεια τώρα θέμα να δώσουμε σε αυτά τα ευρήματα. Έχουμε ένα εσωτερικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο με ε, λεπτομερή ανάλυση. Είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης τώρα με τους ενδιαφερμένους του χρόνου ε, σχεδιάζουμε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών και για εθάρρυνση των κρατών μελών να χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο για να λάβουν δράση. Εδώ σας δείχνω που μπορείτε να βρείτε περισσότερη πληροφόρηση σε αυτό το link. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θα έχετε. Uh, well, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου, λέει ο πρόεδρος. Ε, πραγματικά προσφέρετε τροφή για σκέψη με την παρουσίασή σας για τόσα πολλά πράγματα που κάνουμε. Άλλωστε θα να συντάξουμε έκθεση. Και μας προσφέρατε πολύ υλικό αναφοράς. το οποίο θα εξετάσουμε. Μας μένουν λίγα λεπτά. Ευχαρίστως λοιπόν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Δεκάμπος πρώτος, ο κύριος Ροσφόρ επίσης. Α, βλέπω ότι έχετε ήδη γράψει ε, τα ονόματα. Ροσφόρ, ε, Μόζε, Κάμπος. Άλλος κανείς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την μελέτη. Με συνάρπασε πραγματικά. Βλέπω ότι λειτουργεί και καλά η σχέση συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωστάτ. Με μια λέξη γιατί θα πρέπει να επανέλθουμε και πολλές φορές μάλιστα στα συμπεράσματα της μελέτης, η ιδέα του να καταστούν υπεύθυνοι οι καταναλωτές μου φαίνεται σωστή στρατηγική ουσίας. Ο καταναλωτής θα πρέπει να αναλάβει δράση, να κάνει τις επιλογές του, να μην είναι παθητικό ε, υποκείμενο, ούτε να του προσφέρουμε μασημένη τροφή. Εξάλλου, ωστόσο, θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς ότι η λύση των προβλημάτων περιορίζεται μονάχα στην πλευρά του καταναλωτού. Ε, να γίνει υπεύθυνο καταναλωτή σημαίνει ότι πρέπει να γίνει υπεύθυνοι όλοι οι φορεί τη αγορά. Επανερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το θέμα δηλαδή τη εκπαίδευση της εκπαίδευσης στην κατανάλωση, κάτι το οποίο μαθαίνεται δηλαδή, δηλαδή να γνωρίζει κανείς το επιτόκιο ενός δανείου, πρέπει να μπαίνει στους μαθηματικούς υπολογισμούς που να μπορούν να εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν λοιπόν και πράγματα τα οποία αφορούν τις επιχειρήσεις. Είναι αυτονόητο ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η παρουσίαση ε, ακολουθεί την προηγούμενη. Είδαμε ότι όσο πιο ε, ε, περίπλοκη γίνεται η διαδικασία, τόσο λιγότερες προφορίες παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών στους καταναλωτές. Ακόμα και, αν ο, και ο πρόεδρος μας ε, λαμβάνει ένα SMS που του λέει ποια είναι η τιμή μεταφοράς δεδομένων, πάλι είναι ε, μερική μονάχα η ενημέρωση, διότι δεν γνωρίζει τον όγκο των δεδομένων που θα λάβει. Έχουμε επίσης και μια ευθύνη συλλογικές δημόσιες αρχές δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα λογότυπα για παράδειγμα. Όταν βλέπουμε το θέμα των λογοτύπων, κάτι που ε, υποπίπτει στην αντίληψή μου είναι ότι στην πραγματικότητα ο καταναλωτής μπορεί να κάνει μια καλή επιλογή ή μια άσχημη επιλογή και κυρίως αναφέρομαι στην ε, διαφάνεια 19, ανάλογα με την ικανότητα που έχει το πρόσωπο αυτό, να είναι κατά κάποιο τρόπο αυθόρμητος. Υπάρχουν δηλαδή κάποια λογότυπα τα οποία είναι αυτονόητα και κάποια άλλα που είναι όχι. Για παράδειγμα, ε, ο κίνδυνος είναι κάτι τι, που είναι ένα μεγάλο χ. Ε, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει αμέσως ο καταναλωτής. Από την άλλη μεριά, το ΣΕ, ε, το CE, δεν είναι αυτονόητο. Να λοιπόν δύο λογότυπα τα οποία είναι Ε, μπορεί να είναι και παραπλανητικό, διότι θεωρεί ο καταναλωτή ότι πρόκειται για προϊόν Ευρωπαϊκή παραγωγή. ενώ δεν είναι αυτό. Το ίδιο για την ανακύκλωση. Και αυτό είναι ένα λογότυπο το οποίο είναι κάπου αυτονόητο γιατί δίνει ένα κύκλο που ε, ανανεώνεται κτλ. Αυτά όμω μα αφορούν όλου. Όλοι μαζί λοιπόν, δηλαδή επιχειρήσει, καταναλωτέ, ε, δημόσιε αρχέ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση προ την κατεύθυνση αυτή. Κύριε Σαρλ σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Για μένα είναι άσχημα τα νέα αυτά. Εγώ νόμιζα ότι οι καταναλωτές είχαν περισσότερες γνώσεις για πολλά πράγματα. Και με την τελευταία συζήτηση που κάναμε για την περιαγωγή και τα κινητά τηλέφωνα θα έπρεπε να υπάρχει μια εφαρμογή για τα εφή τηλέφωνα που να επιτρέπει στους ανθρώπους να βλέπουν ποιο είναι το κόστος των διαφόρων πραγμάτων που αγοράζουν. Τέλος, θα ήθελα να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η πρώτη της αντίδραση σε αυτή τη μελέτη. Σκεφτήκατε ότι πρέπει να τα λάβουμε τα πράγματα αυτά υπόψη όταν θεσπίζουμε νομοθεσία στον χώρο της προστασίας του καταναλωτού. Για να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα και ε, δύναμη στους καταναλωτές χρειαζόμαστε βεβαίως περισσότερη παιδεία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται ε, να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και οι επιχειρήσεις και οι αρχές, η εποπτεία των αγορών κτλ. Ίσως χρειάζεται λοιπόν μια συνολικά νέα προσέγγιση της σχέσης αυτής στην Ένωση. Γιατί δεν πιστεύω ότι να δοθεί δύναμη στους καταναλωτές αρκεί. Αναμένουμε βέβαια μια νέα στρατηγική προστασία των καταναλωτών. Θα το εξετάσουμε ίσως βέβαια το θέμα αυτό και νωρίτερα. Ο κύριος Δεκάμπος. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι οι καταναλωτές. Αυτό απορρέει από τη μελέτη και από την παρούσα η οικονομική κρίση, δηλαδή οι καταναλωτές θα γίνουν πιο οξυδερκείς λόγω οικονομικής ε, κρίσης. Έτσι θα γίνουν τα ποιοτικά άλματα. Για μένα τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά καταθλιπτικά, όπως είπε και η Κρίστελ, αλλά και καταστροφικά, αποθαρρυντικά. Γιατί μιλάμε για την Ευρώπη των καταναλωτών, η οποία στην ουσία δεν υφίσταται. Αυτό που με απασχολεί είναι το λογότυπο ναι. CE. Πώς δεν γίνεται κατανοητό. Μόνο το 25% το αναγνωρίζει και έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μεγάλη παραχάραξη αυτού του λογοτύπου CE. Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα έγγραφο για τη στρατηγική σε αυτό το τομέα του χρόνου αλλά τι σκέφτεται η Κομισιόν για το λογότυπο ΣΥΗ, το οποίο δεν είναι αναγνωρίσιμο τελικά από τους καταναλωτές. Θα πρέπει να σας πω και εγώ τα εξή. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι αυτό είναι πρόκληση για μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε ως Επιτροπή με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη γιατί μόλις πέρασε το, ένα πακέτο τουλάχιστον δικαιωμάτων του καταναλωτή. Εάν έχουν δικαιώματα και δεν τα ασκούν οι καταναλωτές, τότε χάνουμε χρόνο. Και αυτό σχετίζεται με πολλά ζητήματα που μας απασχόλησαν. Μιλάμε για ευρωπαϊκή ρύθμιση, όπως ζητούν πολλά κράτη-μέλη ζητούμε νομοθεσία για τους ε, καταναλωτές, αλλά ε, δεν ξέρουμε πώς ε, λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Επίσης, ως προς την ανάλυση ανακράτος μέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση, δηλαδή να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που διαφοροποιούν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Είναι το επίπεδο δραστηριότητας των ενώσεων των καταναλωτών, των ΜΜΕ. Υπάρχουν θέματα που σχετίζονται γενικότερα με τη ρύθμιση, με το πώς ασκείται, με το πώς γίνεται κατανοητή αυτό αφορά βεβαίως ε, και τις οργανώσεις και τις ενώσεις των ε, καταναλωτών, που είναι πιο δραστήριες και που όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συνεισφορά σας. Ο κύριος, ε, η κυρία Τέιλορ ή ο κύριος Μακόλιβερ μπορούν να λάβουν το λόγο. Βλέπουμε ότι είναι εδώ συμπαγής η, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Δεν έχουμε χρόνο αλλά μπορώ να σας δώσω το λόγο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ και για τις ε, ερωτήσεις και για τα σχόλια σας. Συμφωνώ με τα περισσότερα. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ θεώρησα τα στοιχεία καταθλιπτικά και αναπάντεχα, γιατί θεωρούμε ότι η γνώση είναι μεγαλύτερη, η γνώση των καταναλωτών για αυτά τα θέματα. Δεν λέμε ότι οι καταναλωτές πρέπει να τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Εμείς θα πρέπει να δράσουμε ως ε, ε, καταρτίζοντες πολιτικοί και πολιτικές. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και στη μελλοντική μας στρατηγική για να φτάσουμε σε καλύτερες πολιτικές και νομοθεσία. Ιδιαίτερα ως προς τα λογότυπα, διότι ίσως θα πρέπει να έχουμε καλύτερα ε, λογότυπα, πιο παραστατικά, πιο διαισθητικά, ας το πούμε έτσι. Τώρα ως προς τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών, αυτό μας απασχολεί, θα το ε, μελετήσουμε περαιτέρω μαζί με το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Καταβάλουμε προσπάθειες για να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν και που ορίζουν αυτές τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Good. Okay, well, thank you. Uh, Σε ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος από τη ΣΑΝΚΟ που θέλει το λόγο. Όχι. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Έχουμε τις ε, δύο εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας που είναι πολύ χρήσιμο υλικό και που θα απασχολήσει και τους συντάκτες θα υπάρξει ένα follow-up και θα ήταν σκόπιμο να διανύμουμε και αντίτυπα σε, όλα τα, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τις διαφάνειές σας, τα στοιχεία καθώς και τα έγγραφα εργασίας. Θα τα διανύμει η γραμματεία. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα. Έχουμε συνάντηση συντονιστών καταρχήν στις 3 το υπενθυμίζω στους συντονιστές, άρα η Επιτροπή θα συνέλθει στις 4.30, όπου έχουμε μια άλλη μελέτη για την τελωνιακή επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και έχουμε μία συζήτηση με την Επιτροπή και κλεισμένων των θυρών για την ασφάλεια προϊόντος. Λοιπόν, Περιμένω τους συντονιστές στις 3 ακριβώς εδώ και την Επιτροπή στις 4.30. Θα τα πούμε αργότερα. Ευχαριστώ. Γεια σας.